Okay. Right. Um, let's uh, meeting. Καλημέρα. Να αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Θα αρχίσω με τις ανακοινώσεις της Πρόεδρου μέχρι να καθίσετε. Πρώτα απ' όλα, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Δεν βλέπω να έχει κανείς αντίρρηση. Εγκρίνεται λοιπόν. Ανακοινώσεις της Πρόεδρου. Πρώτον, ενημέρωση όσον αφορά τους τριμερείς διαλόγους για τον ενιαίο μηχανισμό με καθάρισεις. Έχουμε πέμπτη συνάντηση τριμερούς διαλόγου χτες. Από τις 3 μέχρι μετά τις 8 πήγε το βράδυ. Για πρώτη φορά λοιπόν είχαμε μεγάλες συζητήσεις με την ελληνική προεδρία ιδιαίτερα για τη διαδικασία λήψης απόφασης. Πρόκειται για το άρθρο 16 και άλλες, ε, άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τον ε, ενιοφθόν μηχανισμό. Ο επόμενος τριμερής διάλογος θα ανακοινωθεί σύντομα. Την επόμενη εβδομάδα νομίζω στο Στρασβούργο. Τώρα, η οδηγία για τις πληρωμές λογαριασμών. Επίσης είχαμε τον επόμενο τριμερή διάλογο στις 11 Φεβρουαρίου όπου συζητήσαμε την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών και το εύρος εφαρμογής της οδηγίας αυτής. Εκεί επιτέθηκε κάποια μικρή πρόοδος, αλλά χρειάζονται παρετέρω συζητήσεις για να επιτευχθεί συμβιβασμός. Τρίτο τριμερής διάλογος προβλέπεται για τις 26 Φεβρουαρίου και εκεί θα επικεντρωθούμε στις διατάξεις που έχουν να κάνουν με την διαφάνεια αλλά και με τις αρμόδιες αρχές όσον αφορά την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Εδώ μου υπενθυμίζουν ότι υπάρχει και αναβολή ανταλλαγής απόψεων όσον αφορά την διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη. Οι ευρωβουλευτές θα θυμούνται ότι την πέμπτη που μας πέρασε εγώ συμφώνησα, επειδή το ζήτησαν πολύ, να αφήσουμε περισσότερο χρόνο να συζητηθεί αυτό το θέμα. την προηγούμενη εβδομάδα σας έφτασε με το σχέδιο μερίσιας διάταξης. Σήμερα λοιπόν θα γίνει αυτή η ανταλλαγή απόψεων, όμως δύο μέλη του ΕΛΚ μου είπαν ότι δεν βολεύει την ομάδα τους γιατί είναι στην Κρακοβία και συνεδριάζουν εκεί. Και είναι δύο που ζήτησαν να γίνει η συζήτηση αυτή, οπότε ζητούν την επόμενη Δευτέρα στις 24 του μηνός να το συζητήσουμε στο Στρασβούργο και συμφώνησαν. Θα είναι λοιπόν στο σχέδιο ημερήσια διάταξη τη επόμενη Δευτέρα που θα έχουμε και το θέμα της Τρόικα. Τώρα μετά την συνάντηση αυτή έχουμε μια συνάντηση κοινή, Εκόν Λίμπε, για να ψηφίσουμε ένα άλλο κομμάτι για την νομοποίηση παράνομου χρήματος. 12.30 ώρα Δύο ρόφους πιο πάνω, τέσσερα και δύο είναι η αίθουσα. Δεν υπήρχε άλλη στιγμή που να μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ένα μικρό διάλειμμα για καφέ. Okay, um, got the important coffee with uh, Ωραία, με τον καφέ θα συνεχίσουμε καλύτερα. Τώρα, καλωσορίζω εδώ τον πρόεδρο του Eurogroup σε ανταλλαγή απόψεων. Πρόκειται για τον οικονομικό διάλογο. Θα συζητήσουμε διάφορα θέματα μαζί του. Πρόκειται για τις ειδικέ συστάσεις για τις διάφορες χώρες. Για 10 λεπτά σας δίνω το λόγο να μας ενημερώσετε και μετά θα περάσουμε στο γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων. 5 λεπτά δηλαδή. Αν χρησιμοποιήσετε 5 λεπτά για την ερώτησή σας, δεν θα έχετε απάντηση. Αν είναι πιο σύντομη η ερώτησή σας, τότε θα έχετε και απάντηση. Το ίδιο ισχύει και από εδώ. Αν δεν εξαντληθεί το πεντάλεπτο μπορείτε να έχετε και δεύτερο γύρο στην ερώτησή σας. Και εδώ μου λένε ότι πρόκειται και για τα προγράμματα μικροοικονομικής προσαρμογής. Λάθο λάθος το έλεγε η μερίσια διάταξη. Και πρόκειται και για το πρόγραμμα εργασιών εν ώψη της Ερενής Συνόδου. Εν πάση περιπτώσει, 10 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Παρακαλώ κύριε Τέσσελμπλουμ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε. ότι κυρίε και κύριοι, νομίζω ότι και εμεί είχαμε το ίδιο πρόβλημα με το λάθο στην ημερήσια διάταξη. Ω εκ τούτου θα αυτοσχεδιάσω. Το 2014 θα είναι ένα έτος κρίσιμο, πιστεύω, όχι μόνο γιατί θα διεξαχθούν οι ευρωεκλογέ, αλλά γενικά για τη ζώνη του ευρώ, καθώς προσπαθούμε να εδραιώσουμε την οικονομική ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να αναφερθώ και στην κατάσταση όπως την έχουμε τώρα, αλλά και στις προτεραιότητες για το μέλλον. Εν γέννη, η οικονομική κατάσταση για την Ευρωζώνη βελτιώνεται, η πραγματική ανάπτυξη του ΑΕΠ επανέρχεται στο, θετικά, στο θετικό πρόσημο τα τελευταία τρία τρίμηνα του 2013 και η οικονομική εμπιστοσύνη βελτιώνεται. Η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά κατά το 2014 και 2015. Αυτό βεβαίως σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην σταδιακή ενίσχυση της ζήτησης στο, ε, στην Ευρωζώνη και από, την εσωτερική, και από τις εξαγωγές αλλά και από την εσωτερική ζήτηση που αναπτύσσεται οι οικονομικές συνθήκες με τις αρθρωτικές μεταρρυθμίσεις βεβαίως θα ε, υποστηρίξουν αυτή την βελτίωση, την ε, θετική τάση στην ε, ζήτηση. Προβλέπεται έλλειμμα χαμηλότερο του 3% για το 2014 καθώς επανερχόμαστε σε μια σταθερή βάση και από τη Eurostat ακούμε ότι έχουμε το, την πρώτη μείωση από το πρώτο τρίμηνο του 2007 του λόγου σε σχέση με ΑΕΠ από κυβερνητικό, στο κυβερνητικό ε, χρέος, κρατικό χρέος. Για να συνεχίσουμε λοιπόν την ε, ενίσχυση αυτών των πολιτικών σταθεροποίησης, κάναμε τον Νοέμβριο συνεδρία τη Ευρωζώνης, του Eurogroup, για να συνεχίσουμε την προσπάθεια που έχουν ξεκινήσει τα κράτη-μέλη με το TUPAC, ε, το, τη δέσμη δύο νομοθετημάτων. Έχουμε εξετάσει επίσης σχέδια προϋπολογισμών, αυτό το λεγόμενο peer review, ε, ε, εξέταση από τους εταίρους που προβλέπεται και στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει κρίσιμη σημασία σε σχέση βέβαια και με, την, με τα όσα προβλέπει το Σύμφωνο σταθεροποίηση και Ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν αυτό το σύμφωνο το έχουν υπόψη πάντα κατά το σχεδιασμό των, ε, ε, κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών του τα κράτη-μέλη, πάντα οι κυβερνήσεις. Βέβαια κατόπιν αυτού έρχεται και η ώρα της υλοποίησης και της στήριση των ε, προϋπολογισμών αυτών και τα κράτη-μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε κίνδυνος παραβίασης των όρων του προϋπολογισμού ή μη του. Ίσως να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να προχωρήσουν οι διορθωτικές κινήσεις στην Ευρωζώνη, αλλά σε πολλά κράτη-μέλη έχουν ε, επιταχυνθεί οι διαδικασίες, γίνονται πιο ανταγωνιστικές ε, οι αγορές μας, πιο ευέλικτες οι αγορές εργασίας, πιο σύγχρονη δημόσια διοίκηση, μεταρρυθμίσει διαρθρωτικέ αναπτύσσονται σε όλε τι χώρε. Οι διαρθρωτικέ αυτέ μεταρρυθμίσει είναι απαραίτητε για την εξασφάλιση αηφόρου ανάπτυξη, βιώσιμη ανάπτυξη σε όλη την Ευρωζώνη και θα απευθύνω εδώ έκκληση για την πιο συντονισμένη προσέγγιση ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, να αποφύγουμε τις παράπλευρες συνέπειες. Ο τομέας παραδείγματι των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ε, στην Τραπεζική Ένωση είναι μια ε, πρόοδος και μπορούμε αντίστοιχα και σε άλλους τομείς να προχωρήσουμε συντονισμένα στη μεταρρύθμισή τους. Και επίσης θα ήθελα να επαναλάβω προηγούμενη έκκληση ότι η διευκόλυνση της ανταγωνιστικότητας και της ενίσχυσης των μεταρρυθμίσεων θα περνούσε μέσα από πιο θαραλέους στόχους εφόσον και όταν υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στα επιτεύγματα των κρατών εκείνων που έχουν υποφεληθεί ευρωπαϊκών προγραμμάτων, προγραμμάτων της Ευρωζώνης, χάρη σε τεράστιες θυσίες των πολιτών των κρατών αυτών, τα προγράμματα πλέον φέρνουν απτά αποτελέσματα. Από την τελευταία μας ακρόαση η Ιρλανδία βγήκε από το πρόγραμμά της, ύστερα από μια συνολική αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού της τομέα και την υλοποίηση ενός σημαντικού και πολύ φιλόδοξου σχεδίου για την εξηγένωση των δημοσιονομικών. Έχουν επανέλθει σε ομαλά επίπεδα, σε επίπεδα πριν την κρίση τα ομόλογα και οι συνθήκες χρηματοδότησης για τις τράπεζες έχουν εξομαλυνθεί. Η οικονομική ανάκαμψη είναι πολύ ισχυρή δηλαδή. Η Ισπανία επίσης έχει επιτυχώς ολοκληρώσει το πρόγραμμα οικονομικής ε, ενίσχυσης, συνδρομής έχει γίνει μια σημαντική βελτίωση ως προς τον τραπεζικό τομέα και την πρόσβαση στη χρηματοδότηση στην Ισπανία. Οι αρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν προχωρήσει, έχει ε, λάβει χώρα και η δημοσιονομική εξυγίανση με θετική οικονομική ανάπτυξη και βελτιωμένη εμπιστοσύνη στην αγορά για την Ισπανία. Η Πορτογαλία, όπως γνωρίζετε, βαίνει προς το τέλος του προγραμματός της, το οποίο τηρεί τους όρους του πλήρως. Η τελευταία ενδιάμεση έκθεση αποδεικνύει επιτυχία για την Πορτογαλία και ε, ανάπτυξη εξαγωγές με καλά δείγματα ανάκαμψης. Μάλιστα μόλις τώρα το προηγούμενο μήνα η Πορτογαλία έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ε, εξασφάλιση δυνατότητας εισόδου στις αγορές με την έκδοση ομολόγων που είχαν πολύ σημαντική ε, διεθνή ζήτηση. Για την Ελλάδα μπορεί να υπάρχει ακόμα μακρύς δρόμος μπροστά. Ωστόσο είναι πολύ σημαντικές οι ε, σημαντικά τα επιτεύγματα έχει ε, προβλέπεται ότι θα υπάρξει πρωτογενές πλεόνασμα για το 2013. Αυτό μας λέει η κυβέρνηση. Περιμένουμε και τα αποτελέσματα της Eurostat στα τέλη Απριλίου. Το ε, έλλειμμα τρέχουσων συναλλαγών εξαλείφθηκε τα τελευταία τρία χρόνια και ο λόγος χρέους προς το ΑΕΠ. Πιστεύουμε ότι αυτό το χρέος θα αρχίσει να μειώνεται ε, με την παράλληλη οικονομική ανάπτυξη. Η αναθεώρηση για την Ελλάδα πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να ολοκληρωθεί σύντομα μόλις ολοκληρωθούν οι όροι για την τήρηση, τήρηση του προγράμματος. Και από ό,τι φαίνεται η Τρόικα θα επανέλθει την Κυριακή στην Αθήνα, θα επιστρέψει την Κυριακή. Η Κύπρος έχει ένα πρόγραμμα ε, Προσαρμογή εξυγίανση που βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ακόμη, αλλά έχουν αναλυφθεί σημαντικά μέτρα, αναδιάρθρωση, ανακεφαλαίωση του τραπεζικού ε, τομέα, έχει προχωρήσει σημαντικά και βλέπουμε από την αποστολή ε, αναθεώρηση μελέτη, ότι ήδη η κατάσταση σε σχέση με το 2013 είναι πολύ καλύτερη από ό,τι προβλεπόταν και ο χρηματοπιστωτικός τομέας σταθεροποιείται. Εν όλο, οι πρόσφατες εξελίξεις είναι θετικές επιβεβαιώνουν πιστεύω τη στρατηγική μας και γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε την στρατηγική αυτή στα κύρια στοιχεία τους της. Βεβαίως οι δυσκολίες είναι σημαντικές για τους πολίτες της Ευρώπης και βεβαίως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα υψηλά επίπεδα ανεργίας που θεωρούμε απαράδεκτα, πρέπει να καταφέρουμε καλύτερα αποτελέσματα στις οικονομικές μας επιδόσεις. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και εκεί χρειάζεται περισσότερη ε, επιτάχυνση στο θεματολόγιο. Έχω ακόμα χρόνο, δύο λεπτά. Είναι κρίσιμη σημασία για όλη την Ευρώπη, αλλά ιδιαίτερα και την Ευρωζώνη, να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο το δυναμικό μας για την ανάπτυξη και κύριος στόχος εν προκειμένου είναι να διατηρήσουμε το κοινωνικό μοντέλο, να διαφυλάξουμε το κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης. Το έχω ξαναπεί ότι υπάρχει πολύ περιθώριο για βελτίωση στον χώρο αυτό. Η Τραπεζική Ένωση έχει πολύ μεγάλη σημασία για, το Eurogroup και την Ευρώπη γενικότερα. Έχει κέρια σημασία για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στην οικονομία της Ευρώπης. Όπως γνωρίζετε, ετοιμάζουμε, η καλύτερη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζει τον ε, μηχανισμό εποπτείας με την ε, ε, επιθεώρηση, αναθεώρηση καλύτερα και τα τεστ αντοχής προσδιορίσει προς το παρόν τη μεθοδολογία που θα αξιοποιήσει. Στόχος μας είναι το λειτουργικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σταθεροποιητικού Μηχανισμού με το μέσον RECAP να είναι έτοιμο ε, το Μάρτιο, με την φύση όπως έχουμε συμφωνήσει από τον Ιούνιο πέρσι. Για το SRM ξέρετε ότι προχωράει υπό την ευθύνη της ελληνικής προεδρίας, το ΕΚΟΦΗΝ, ωστόσο μπορούμε να προχωρήσουμε σύντομα ώστε να είμαστε έτοιμοι πριν τον ε, Απρίλιο για τη Σύνοδο του Κοινοβουλίου. Αυτή την εβδομάδα έχουμε ειδική υπουργική συνεδρίαση για το ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης. Είχαμε συνάντηση τη Δευτέρα με τους εμπειρογνώμονες όπου εντοπίστηκαν τα ζητήματα και εξασφαλίστηκε ε, σύγκληση απόψεων σε μια σειρά από σημαντικούς τομείς. Συνεχίζουμε τις προσπάθειες με μια ειδική και πάλι συνάντηση υπουργών το Μάρτιο. Όλοι οι εμπλεκόμενοι δεσμεύονται για ε, εξασφάλιση συμφωνίας μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Αυτά προς το παρόν και σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ που τηρήσατε και το χρόνο σας. Όντως είχαμε τον πρώτο καρποφόρο τριμερή διάλογο χτες. Μετά την απόφαση να επιτρέψουμε στην Ελληνική Προεδρία κάποια ευελιξία. Ήταν κρίμα που δεν έγινε αυτό τέσσερις τριμερείς διαλόγους νωρίτερα. Χρειάστηκε να δουλέψουμε σκληρά. Τώρα δεν ξέρω πότε τον Απρίλιο, αλλά ελπίζω να τα καταφέρουμε. Παρόλο που εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές βέβαια, αλλά θα κρατήσω αισιόδοξη στάση. Εκ μέρους του ΕΛΚ, Παύλος Άλμπα, η πρώτη ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πρόεδρε, συμφωνώ μαζί σας. Πιστεύω και εγώ ότι τα πράγματα πάνε κάπως καλά και βλέπουμε φως στο τέλος του τούνελ. Εμένα με απασχολεί το θέμα των πιστώσεων, διότι εδώ με την πτώση είναι δύσκολο να πετύχουμε σταθεροποίηση οικονομική. Οπότε στην Ευρώπη πώς θα καταφέρουμε να πετύχουμε πιστώσεις που να ρέουν, ιδίως στις χώρες του Νότου της Ευρώπης. Έπειτα για την ε, ανακεφαλοποίηση των τραπεζών από πλευρά του Μέντε. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε κατά πόσο οι προϋποθέσεις, οι συνθήκες είναι σαφείς. Με τους κανόνες που υπάρχουν για τη βοήθεια στις τράπεζες, είχα καταλάβει ότι ήταν σαφείς οι προϋποθέσεις, αλλά τώρα κάποιοι ζητούν να εφαρμοστούν προδιαγραφές της οδηγίας για την ανάκαμψη των τραπεζών. Στο Eurogroup συζητήσατε καθόλου τι συνέπειες θα είχε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ για την... τις δύο ερωτήσεις σας ουσιαστικά. Πρώτα απ' όλα για τη ρευστότητα της πιστώσης που θα θέλαμε να δούμε ξανά να κυκλοφορούν και μέσα και εκτός Ευρώπης για να υποφεληθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει η Τραπεζική Ένωση, πάνω σε αυτό δουλεύουμε κυρίως, γιατί αυτό θα βοηθήσει. Και ξέρετε ότι από τον Νοέμβριο υπάρχουν εξελίσεις. Το δεύτερο στοιχείο κλειδί για να πετύχουμε ξαναπιστώσεις, εντάξει μπορεί να απαντάει ακριβώς στην ερώτησή σας, αλλά είναι η ανάκαμψη. Όσο πιο γρήγορα έχουμε εξελίξεις για τα δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται, τόσο πιο γρήγορα θα έχουμε και πάλι ρευστότητα. Τώρα υπάρχουν θετικά στοιχεία στην οικονομία, αλλά παραμένουν δάνεια που δεν έχουν επιληθεί. Έπειτα, χρειαζόμαστε και κάποιες γραμμές βοήθειας αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, προκειμένου να έχουμε πιστώσεις. Ακόμα και αν οι τράπεζες ακόμα ε, κοιτάνε τι θα κάνουμε τις απώλειές τους και αν δεν είναι ακόμα αρκετά δυνατές, παρόλα αυτά πρέπει να μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το ECP σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για προγράμματα από την ε, Κεντρική Τράπεζα, Σύλλομη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ναι, και εξετάζονται διάφορες δυνατότητες. Οι χώρες λοιπόν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους μέσα. Βέβαια έχει γίνει πολλή δουλειά, αλλά πρόκειται για γραμμές βοήθειας, για να το πω έτσι. Δεν πρέπει να υπάρχει κατακαιρματισμό τη δημοσιονομική αγορά στην Ευρώπη. Πρέπει να υπάρχει ρευστότητα και, προ... και πιστώσεις και προς τι επιχειρήσει και γενικότερα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τώρα για τη δεύτερη ερώτησή σας, κατά πόσο οι προϋποθέσεις είναι ξεκάθαρες. Δεν έχουμε τελειώσει με την πρότασή μας. Υπάρχει μια πολιτική απόφαση από τον Ιούνιο που μας πέρασε για τα κυρία στοιχεία. Οι προϋποθέσεις ήταν σαφείς, δηλαδή πρέπει να πρόκειται για τράπεζες οι οποίες είναι βιώσιμες, τράπεζες οι οποίες συστημικά να έχουν τη σημασία τους, δηλαδή ο ενιαίος ε, μηχανισμός ε, επίλυσης εκαθάρισης δεν θα βοηθήσει τράπεζες οι οποίες έτσι κι αλλιώ δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν. Αν οι χώρες τώρα μπορούν οι ίδιες να βοηθήσουν τις τράπεζές τους, τότε πρέπει να το κάνουν, αλλιώς βεβαίως θα υπάρχει αυτή η βοήθεια μόλις έχουμε το recap. Μόλις έχουμε την ε, ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Και βέβαια πρέπει να προβλέψουμε και το in-bail, έτσι, την διάσωση με ίδια μέσα. Τώρα συζητάμε πόσο μακριά θα πάει αυτό, πόσο καλά θα λειτουργήσει. Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο ακόμα συζητάμε. τότε μόνο θα ξέρουμε τις τελικές λεπτομέρειες. Ακόμα δεν τις έχουμε. Πολλές προϋποθέσεις είναι σαφείς, σας τις είπα, αλλά υπάρχουν και κάποιες που ακόμα συζητιόνται. Το καυτό θέμα είναι οι ομολογιούχοι. Εξαρτάται από τον ισολογισμό της τράπεζας. Γιατί αν πείτε ότι πρέπει να είναι 8% bail σας είπα, ακόμα το συζητάμε, έτσι δεν ξέρω ποιο θα είναι το τελικό ποσοστό, αλλά αν έχετε ένα 8% bail-in, τότε μπορεί να αφορά και τους ομολογιούχους. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η Άννη Ποδηματά, εκ των Σοσιαλιστών, παρακαλώ. Thank you, Sharon, κύριε Πρόεδρε. Ε, συμφωνώ μαζί σας ότι έχουν υπάρξει τα πρώτα σημάδια οικονομικής ανάκαμψης ε, ωστόσο, όπως επισημάνατε και εσείς, επισημαίνει και υπογραμμίζει και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι πολύ εύθραυστα ακόμα αυτά τα σημάδια της ανάκαμψης της οικονομίας και υποθέτω ότι αυτή η ανάκαμψη δεν είναι αρκετή για να κατευνάσει τις ανησυχίες που εξακολουθούν να υπάρχουν για την ε, βιωσιμότητα, ε, για τα επίπεδα του χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στην Ευρωζώνη. Επειδή συζητήσατε λοιπόν και στο Eurogroup και στο ECOFIN για την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης, επειδή υπογραμμίζουμε συνέχεια στα λόγια την ανάγκη μιας φιλικής προς την ανάπτυξη δημοσιονομικής προσαρμογής, πέρσι το υπογραμμίσαμε, δεν τη βλέπουμε να συνοδεύεται με πράξεις. Ταυτοχρόνως έχουμε πρωτόγνωρα επίπεδα ανεργίας στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη, ιδιαίτερα στην Ελλάδα και στην Ισπανία, το 1 τρίτο του ενεργού πληθυσμού ε, βρίσκεται σε ανεργία. Θέλω να σας ρωτήσω ε, εάν είστε ικανοποιημένος από αυτά που γίνονται σε αυτό το επίπεδο για να σταθεροποιήσουμε και να ενισχύσουμε την ανάκαμψη και να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πρωτόγνωρα επίπεδα ανεργίας. Ενώ ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην, ε, Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε, είπατε και σωστά ότι κατά τις εκτιμήσεις τις με των ελληνικών αρχών και τη κυβέρνηση θα υπάρξει νωρίτερα από το αναμενόμενο ένα πρωτογενές πλεόνασμα που βεβαίω αναμένουμε να επικυρωθεί τον Απρίλιο από την Eurostat. Ε, θέλω να σας ρωτήσω, ε, στη βάση αυτού του, ε, αυτής της επικύρωσης των στοιχείων από την Eurostat, ποιες είναι οι εναλλακτικές που εξετάζετε για να ε, ε, λυθεί το θέμα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Διότι όσο αυτό δεν λύνεται κύριε Πρόεδρε, τόσο υπάρχει ανασφάλεια και στους επενδυτές, εγχώριους και ξένους και άρα καθυστερεί και η ανάκαμψη γιατί παρατείνεται το κλίμα βεβαιότητας. Και τελευταίο, εάν στις εναλλακτικέ που θα εξετάσετε για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους περιλαμβάνεται ή θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και η αναδρομική απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, σε συνέχεια και της ε, ερώτησης του Πάμπλο. Συζητήσατε την Τρίτη, ε, Υπουργή για αυτό το θέμα και θέλω να σας ρωτήσω αν είναι ε, μία από τις λύσεις που θα μπορούσατε να εξετάσετε. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Η πρώτη ερώτηση ήταν κατά πόσο είμαι ικανοποιημένος. Όχι, δεν είμαι. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να είναι ικανοποιημένος. Το επίπεδο βέβαια ανάπτυξης βελτιώνεται. Περισσότερο μάλιστα από ό,τι είχαμε προβλέψει οικονομική ανάπτυξη. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος. Σίγουρα δεν είμαι ικανοποιημένος με τα υψηλά επίπεδα ανεργίας που υπάρχουν σε πολλές χώρες και δεν λένε να μειωθούν. Βέβαια, βγαίνοντα από μια κρίση, χρειάζεται χρόνος μέχρι η ανεργία να αρχίσει να μειώνεται. Αλλά δεν είμαι ικανοποιημένο. Και γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι πρέπει τα επόμενα χρόνια να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι στην ημερήσια διάταξή μας, στους στόχους μας, για να κάνουμε την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική. Βέβαια, υπάρχει δυνατότητα Άλλοι λένε δεν μπορεί η Ευρώπη να αναπτυχθεί περισσότερο από μισό της εκατό. Όχι, υπάρχει και η ανάλυση αναχώρα δείχνει ότι αν γίνουν τα σωστά πράγματα, αν δηλαδή γίνουν διορθώσει στην οικονομία, στον τρόπο που λειτουργεί η διακυβέρνηση, οι αγορέ κτλ. Υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερη ανάπτυξη και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την πετύχουμε αυτή την οικονομική ανάπτυξη. Για την Ελλάδα πιο συγκεκριμένα. Όπως γνωρίζετε, το Eurogroup τον Νοέμβριο του 2012 είπε ότι όταν υπάρξει πρωτογενές πλεόνασμα και από ό,τι φαίνεται αυτό θα φανεί τον Απρίλιο από τα νούμερα και εφόσον η Ελλάδα έχει καλύψει τις προϋποθέσεις του προγράμματος, τότε θα κοιτάξουμε τη βιωσιμότητα του χρέους πιο μακροπρόθεσμα. Αυτό συμπίπτει με την απόφαση που πρέπει να ληφθεί το δεύτερο εξάμενο της χρονιάς αυτής, για το μέλλον του ελληνικού προγράμματος. Όπως ξέρετε το τρέχον πρόγραμμα λύγει στα τέλη της χρονιάς και θα πρέπει να αξιολογήσουμε το δεύτερο εξάμεινο της χρονιάς αυτής κατά πόσο χρειάζεται νέο πρόγραμμα και τι μορφή θα έχει αυτό. Υπάρχουν κάποιες αισιόδοξε φωνές από την Ελλάδα που λένε ότι ίσως δεν θα χρειαστεί καθόλου. Μακάρι. Θα δούμε όμως, βάσει των στοιχείων που θα έχουμε μέσα στη χρονιά και ανάλογα θα είναι και αποφάσεις που θα πάρουμε το δεύτερο εξάμεινο για το μέλλον. Τώρα για εναλλακτικές αναφερθήκατε στις τράπεζες. Το τραπεζικό τμήμα του ελληνικού προγράμματος εφαρμόζεται. Υπάρχουν ε, οι δοκιμές αντοχής για την ποιότητα και τα λοιπά σε ελληνικές τράπεζες. 10 εκατομμύρια είναι στην πάντα για αυτόν ακριβώς το σκοπό, για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και θα δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό. Τότε θα υπάρξουν νέα χρήματα να μπουν στις τράπεζες για να υπάρξει ανακεφαλοποίησή τους. Πάντως για όλες τις τράπεζες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα τις ξαναπεράσει από τη διαδικασία και η EBA θα κάνουν τις δοκιμές αντοχής και στα τέλη της χρονιάς θα ξέρουμε ακριβώς που βρισκόμαστε. Είναι ζωτική σημασία για την ανάκαμψη και στην Ελλάδα να έχει ισχυρέ τράπεζες ώστε να μπορούν να χρηματοδοτούν νέες επιχειρήσεις, να δώσουν νέες δυνατότητες στις επιχειρήσεις και αυτό είναι μέρος της προσέγγισής μας. Όσον αφορά το μέλλον, νομίζω ότι είναι ζωτική σημασία, αλλά αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, έχει να κάνει με την στρατηγική μας γενικά. Υπογραμμίζουμε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αναπόφευκτα, τη δημοσιονομική πτυχή, τα σταθερά δημοσιονομικά ώστε να μπορούν οι χώρες να επαναχρηματοδοτούνται στο μέλλον. Τώρα, αυτό πρέπει βέβαια να το μεταφέρουμε λιγάκι και στις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κάνουν οι χώρες. Πάντα με την Ελλάδα υπάρχουν ερωτήσεις, ε, απάντηση δεν είναι απλή, πολλά πράγματα γίνονται αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα. Σιλβή τώρα, από τους φιλελεύθερους. Σας ευχαριστώ και ε, Υπουργέ που είστε μαζί μας. Ε, θα συνεχίσω στα γαλλικά αν δεν σας πειράζει. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και σας ευχαριστώ που μας δώσατε την ευκαιρία ως ε, ε, συντάκτες του ψηφίσματος να έρθουμε να συζητήσουμε με τους υπουργού της προάλλης. Ήταν μια σημαντική εμπειρία για να δούμε τις δυσκολίες που έχετε να συμφωνήσετε, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει επίσης να κατανοήσουμε καλύτερα τις αμφιβολίες ημέν των δε. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε κάτι απλό το οποίο ζητάμε. Δηλαδή μια ε, νομική μελέτη εις βάθος που θα μας εξηγήσει γιατί πρέπει να κάνουμε εξαίρεση στις αρχές σύμφωνα με τις οποίες ε, ε, συντάσσεται η νομοθεσία σε συναπόφαση με το Συμβούλιο. Είναι ένα θέμα το οποίο θίγεται. Είχαμε χθε μια βιντεοδιάσκεψη με τον Bundestag, κάτι το οποίο ρωτούν οι Γερμανοί βουλευτέ, του οποίου σεβόμαστε απολύτω, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε αν επί τη ουσία είναι νομική διεκδίκηση, επί τη οποία μπορούμε να εργαστούμε, αν πρόκειται για πολιτική φύση διεκδίκηση, διότι είναι πολύ περίπλοκο να γίνουν όλα αυτά με το, με το Κοινοβούλιο. Σας καλώ λοιπόν και γνωρίζω τον επικοδομητικό ρόλο που έχετε παίξει στο πλαίσιο του Eurogroup για να πιέσετε του τους ε, εταίρους σας να ενεργήσουν, να δράσουν, να προσεγγίσουν το Κοινοβούλιο, αλλά όπως είπε και η Πρόεδρός μας, ο πρώτος τριμερής διάλογος που είχαμε την αίσθηση πως κάπως, πως οι συνομιλητές μας είχαν ε, τη διάθεση να συνομιλήσουν, ήταν χτες. Χάσαμε δύο μήνες και είναι κρίμα. Ε, η συναπόφαση δεν σημαίνει ότι το Συμβούλιο αποφασίζει και το Κοινοβούλιο απλά επικυρώνει, όπως λένε. Ε, τώρα, έχω και κάποια σχόλια επί της ουσίας. Εχθές είδε ένα διασκεδαστικό έγγραφο, πολύ διασκεδαστικό μάλιστα, χωρίς να θέλω να σας πειράξω, που λέει ότι η απόφαση του Συμβουλίου θα μπορούσε να ληφθεί σε ένα Σαββατοκύριακο. Αλλά εγώ ε, δέχομαι αμέσω την έννοια του Σαββατοκύριακου, κύριε Υπουργέ, γιατί το Σαββατοκύριακο ξεκινά την Παρασκευή το απόγευμα και τελειώνει την Τετάρτη το μεσημέρι, την επόμενη Τετάρτη το μεσημέρι. Ωραία θα ήταν όμως πώς θα ξεκινήσουμε μια τόσο περίπλοκη διαδικασία που δεν ξέρουμε πόσες μέρες θα μας χρειαστεί να λάβουμε μια απόφαση. Είναι προφανές ότι αν μια τράπεζα πρέπει να κλείσει μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα το πρωί πρέπει να έχει ληφθεί απόφαση. Και το γεγονός επίσης ότι οι αρχές αναμεγνύονται τόσο πολύ με το Συμβούλιο της Επιτροπής ε, ε, καθάρισης και τα λοιπά. Πώς θα μπορέσουμε να αναλάβουμε με τέτοια ευθύνη, πώς θα έχουμε έλεγχο από τη στιγμή που δεν ξέρουμε ακριβώς εμείς ποια θα είναι η αρχή η οποία θα φέρει την ευθύνη για μια τόσο σοβαρή απόφαση όπως είναι το κλείσιμο μιας τράπεζας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Δεν θα ήθελα να μπω σε υπερβολικές λεπτομέρειες ε, γιατί όπως ξέρουμε θα το διαπραγματευτούμε όλα αυτά και όπως είπα το SRM είναι η ευθύνη της ε, ελληνικής προεδρίας. Εγώ προεδρεύω στην διακυβερνητική ε, και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις αντιρρήσεις του κοινοβουλίου σε αυτό το οικοδόμημα. Το ερώτημά σας είναι, είναι πολιτικό ή νομικό το ζήτημα. Σίγουρα είναι νομικό θέμα όχι μόνο από ευρωπαϊκή νομική οπτική, αλλά και από πλευράς κάποιων εθνικών συνταγματικών νομικών πτυχών που το καθιστούν το θέμα εξαιρετικά περίπλοκο. Για να είμαι ειλικρινής λοιπόν, η διακυβερνητική συμφωνία θα είναι κομμάτι του συνόλου του SRM, αλλά ξέρω πως πιστεύετε κάτι το διαφορετικό εσείς. Πάντως έτσι έχουν τα πράγματα και θα πρέπει να κάνουμε, πιστεύω ότι μπορούμε, και αυτή ήταν η δεύτερη σας παρατήρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ένα Σαββατοκύριακο θα τελειώνει στις 8 η ώρα το βράδυ της Κυριακής και ότι θα έχουμε αποφάσεις που θα είναι αποτελε... μάλλον μια διαδικασία λήψη αποφάσεων αποτελεσματική. Ε, και ταχεία. Αυτή ήταν μια από τις πρώτες αρχές που ε, ε, ανέφερε η κυρία Φερέρα όταν ήταν στην ε, συνεδρίασή μας τη Δευτέρα το βράδυ. Ότι δηλαδή θα πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις γρήγορα όσον αφορά την εκαθάριση τραπεζών. Αυτό εξετάζουμε λοιπόν που είναι δυνατόν να γίνει όλη αυτή η διαδικασία πιο αποτελεσματική και πιο ταχεία. Αναγνωρίζω λοιπόν ότι υπάρχει θέμα εδώ και ότι υπάρχει χώρος για βελτίωση, όπως είπαν και οι συνάδελφοι ήδη. Σας ευχαριστώ και τώρα περνάμε στους πράσινους. Μπας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ Ντάισελμπλουμ. Έχω τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, όσον αφορά την ε, εποπτεία. Ο κύριος Φαντρομπάλ είχε υποσχεθεί ότι θα υπάρξει κοινοβουλευτική εποπτεία και θα υπάρξει διαθεσμική συμφωνία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Eurogroup. Δύο χρόνια μετά δεν έγινε. Πότε θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την διοργανική αυτή συμφωνία ώστε να υπάρξει μεγαλύτερος κοινοβουλευτικός έλεγχος στον ενίο αυτόν μηχανισμό εξηγένσης. Δεύτερον, την ε, Δευτέρα που μας πέρασε είχαμε μια επιτυχία με 2 εκατομμύρια για την πρωτοβουλία πολιτών που δεν θέλουν τη ιδιωτικοποίηση του νερού. Μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, εσείς το 2013 το Δεκέμβριο αναφερθήκατε στην Ελλάδα και είπατε ότι απαιτείται ιδιωτικοποίηση του νερού στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν υπάρχει λόγος να πιεστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εσείς λοιπόν τι θα κάνετε τώρα ώστε να πετύχει η πρωτοβουλία αυτή πολιτών και η Τρόικα να μην επιβάλλει την ιδιωτικοποίηση του νερού στην Ελλάδα. Τρίτη ερώτηση. Είπατε ότι είναι απαράδεκτη ενέργεια; το είπατε πριν από λίγο. Ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε τέτοια ανεργία. Οπότε αναρωτιέμαι τι εννοείτε γιατί αυτή τη βδομάδα το Eurogroup και το ECOFIN συζήτησαν για τους κοινωνικούς δείκτες. Ότι πρέπει να έχουμε περισσότερη κοινωνική Ευρώπη και το δικό σας ε, κόμμα στο πρόγραμμά του το λέει αυτό. Αλλά τα συμπεράσματα του ECOFIN της Τρίτης με τους δείκτες που θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για μια ευρύτερη κατανόηση των κοινωνικών εξελίξεων. Τι σημαίνει αυτό. Να δούμε αν θα είναι καλά τα πράγματα ή όχι. Μα τι θα κάνετε ώστε οι κοινωνικοί δείκτες να επιβληθούν και όχι μόνο για λόγους κατανόησης, αλλά για να αλλάξει και κάτι. Αυτά μετά τα συμπεράσματα του ΕΚΟΦΗΝ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω στα αγγλικά. Τρεις ερωτήσεις πρώτο για την ε, δημοκρατική λογοδοσία του ενιαίου μηχανισμού σταθεροποίησης. Όπως ξέρετε είναι διακυβερνητικός ο ESM. Ως εκ τούτου οι υπουργοί που ταυτόχρονα έχουν και την ευθύνη απευθύνονται στα εθνικά τους κοινοβούλια, λογοδοτούν σε αυτά. Και αν, αν γνωρίζω καλά και ο, προκατοχός μου κύριος Γιούνκερ είχε αποστείλει στο κοινοβούλιο σα επιστολή λέγοντας ότι θα ενημερώνετε τακτικά το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βεβαίω πάντα είμαστε στη διάθεσή σα, είμαστε έτοιμοι και ικανοί να προσφέρουμε αυτή την ε, πληροφόρηση. Έχει αποστελεί νομίζω στον υποφαινόμενο τον κύριο Ρέγκλινγκ η σχετική πρόσκληση για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Πάντω, αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, μπορείτε να την υποβάλλετε τώρα. Γι' αυτό είμαι εδώ εγώ. Γιατί να τα περιπλέκουμε τα πράγματα. Εδώ είμαι, ρωτήστε μου ό,τι θέλετε. Αυτή είναι η απλή λύση για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθεροποίηση. για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Τα συμπεράσματα στα οποία αναφέρεστε λέγουν ότι η λέξη required απαιτείται για τον εξή λόγο, ότι ήταν κομμάτι του προγράμματος ιδιωτικοποίησης των πόρων στην Ελλάδα. Κανείς δεν υποχρέωσε την Ελλάδα να βάλει την εταιρεία υδάτων της μέσα στο πρόγραμμα για την ιδιωτικοποίηση αλλά αποτελεί κομμάτι των σημαντικών προσπαθειών για την ιδιωτικοποίηση των δημοσίων εταιριών της Ελλάδας. Κομμάτι του προγράμματος για τον περιορισμό του χρέους για την εξυγίανση των δημοσιονομικών της Ελλάδας. Αυτό ήταν ένα μέρος, η ιδιωτικοποίηση. Οι επιχειρήσεις οι οποίες επελέγει σαν και μπήκαν στο πακέτο των ιδιωτικοποίησεων είναι η υπόθεση της Ελλάδας και όχι της Ευρώπης. Κάποιοι επιλέγουν να, να πούν ότι η Ευρώπη ευθύνεται για τα πάντα, αλλά δεν είναι αλήθεια. Κοινωνικοί δείκτες και στόχοι αυτών. Η διατύπωση συμφωνώ ότι δεν φαίνεται ιδιαίτερα φιλόδοξη μόνο αντίληψη, κατανόηση κτλ. Αλλά για να σας εξηγήσω, ο λόγος που θέλουμε να καταλαβαίνουμε τις κοινωνικές επιπτώσεις αυτών που πράττουμε είναι για να βοηθηθούμε να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις στη μακροοικονομική μας πολιτική. Επομένως παρακαλώ να μην παρερμηνεύσετε τον όρο soul purpose of understanding, μόνος λόγος ή κατανόηση ή αντίληψη. Πρέπει να είμαστε θέση να αντιλαμβανόμαστε ποιες είναι οι κοινωνικές συνέπειες για να τις λαμβάνουμε υπόψη. Βλέπω ότι έχω 50 δευτερόλεπτα, λέει ο κύριο Eichhout. Μια και μου δώσατε την ευκαιρία για το πρώτο θέμα. Ξέρετε ότι το Ολλανδικό Κοινοβούλιο δεν έχει δικαίωμα άρνηση κυρία για οποιαδήποτε πληρωμή σε σχέση με το μηχανισμό σταθεροποίηση. ενώ το Γερμανικό έχει. Άρα έχουμε πρόβλημα νομοποίησης, ε, δημοκρατικής νομοποίηση στον ESM. Ο Φαν Ρόμπο είχε υποσχεθεί ότι θα υπάρξει ένα ε, τρόπο να ρυθμιστεί το θέμα αυτό. Ερωτώ λοιπόν, και μάλιστα πριν από εσά πριν να λάβετε εσεί καθήκατα, ερωτώ λοιπόν, πέραν των ωραίων συζητήσεων που κάνουμε, συγκεκριμένα τι μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε τη δημοκρατία δεν ξέρω, λέει ο κύριος Δάισελμπλουμ, προλαβαίνω να απαντήσω. Η απάντηση ήταν η εξής. Εάν πιστεύετε ότι το Ολλανδικό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να επιτρέψει προγράμματα και πληρωμές σχετικές με προγράμματα για χώρες ε, της Ευρωζώνης να περάσουν, τότε απαντάστε. Διότι πολλές συζητήσεις γίνονται στο, στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο που είναι σχετικές με το θεμετολόγιο ε, με τα θέματα προσυζήτηση στο Eurogroup, στην Ευρωζώνη. Και αν η πλειονότητα των βουλευτών του Ολλανδικού Κοινοβουλίου πει «Κύριε Υπουργέ, δεν συμφωνούμε με την τάδε πληρωμή, με το τάδε ποσό», ε, τότε προφανώς έχω πρόβλημα. Υπάρχει λογοδοσία, υπάρχει σαφέστατα υποχρέωση λογοδοσίας, τόσο στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο, όσο και στο Γερμανικό, αλλά και σε πολλά άλλα. Καλώς λέει ο Πρόεδρος, αργήσαμε λίγο ε, να βάλουμε το χρονόμετρο να δουλεύει. Τέλος πάντων χρήσιμο ήταν και αυτό. Γιούργεν. Ευχαριστώ, Σάουρον, και θα μιλήσω γερμανικά. Δύο ερωτήσει. Με παρακολουθείτε? Ωραία. Λοιπόν, η πρώτη μου ερώτηση. Έχει να κάνει με την απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Καρσούης ε, για τον μηχανισμό εξυγίανσης και το είναι Ευρωζώνη και το δεύτερο για την Ελλάδα. Η κυρία Ποδηματά επιβεβαιώνει και από πλευρά τη ότι έχουμε κάποια πρώτα θετικά βήματα. Ωστόσο, εχθέ ο Υπουργό Σόιμπλε τη Γερμανία ξεκίνησε, προκάλεσε διάλογο λέγοντα ότι η Ελλάδα έχει πτωχεύσει και ότι χρειάζεται περικοπή, ε, ανάταξη, περικοπή του χρέους η Ελλάδα. Πώς λοιπόν, κούρεμα να το πω έτσι, Πώς λοιπόν ε, βλέπετε εσείς την κατάσταση όταν λέτε στην αρχή της ομιλίας σας όπως και η κυρία Ποδηματά ότι η Ελλάδα πάει καλύτερα, χρειάζεται αυτός ο διάλογος ο δημόσιος ή όχι. Απάντηση. Πρώτον, για το Σταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας. Παρακολουθώ την ανάλυση της απόφασης αυτής, η οποία γίνεται αντικείμενο πολλαπλών συζητήσεων και ερμηνεών. Εγώ παραμένω στο γεγονότο ότι δηλαδή παραπέμπουν το ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και άρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε από εκεί τι θα προκύψει. Το μόνο που μπορώ να πω όμως είναι πως λυπούμε που δεν έχει ολοκληρωθεί ο διάλογος για το μέσον αυτό το οποίο έχει αποδειχθεί τόσο χρήσιμο όσο και αν δεν το έχουμε ε, αξιοποιήσει ουσιαστικά έχει φέρει με την ύπαρξή του την σταθεροποίηση στην Ευρώπη. Και πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να το χρησιμοποιούμε, αλλά όπως και να και εγώ περιμένω την απόφαση του δικαστηρίου και οποιαδήποτε βέβαια άλλη ανάλυση των συνεπειών ή ε, οτιδήποτε προκύψει από το παραπεμπτικό αυτό βούλευμα για προδικαστικό του δικαστηρίου της Καλσούης. Για την Ελλάδα δεν άκουσα να λέει κανείς ότι έχει πτωχεύσει. Με εχτές, ε, εχτές ένα μεγάλο άρθρο στη Handelsblatt της Γερμανίας, γερμανική εφημερίδα που ονομάζεται Handelsblatt και είναι σημαντική οικονομική εφημερίδα, υπήρχε αυτή η αναφορά. Καλώ λέει ο κύριο Τάσιμπλουμ, αλλά δεν μπορώ να. Το μόνο μπορώ να σα πω είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει πτωχεύσει ξεφεύγει από την κρίση σιγά σιγά, έχει να επιδείξει θετικό ε, πρωτογενές αποτέλεσμα, πρωτογενές πλεόνασμα δηλαδή, δεν θέλω να συζητήσω σε όρους που να αναθεωρούν το που βρισκόμαστε. Αλλά πολύ ευχαριστώ θα διαβάσω το άρθρο αυτό της Handelsblatt, την οποία γνωρίζω ως εφημερίδα, αλλά δεν είχα την ευκαιρία να αναγνώσω το εν λόγω άρθρο. Ο κύριος Κλούτε θέλει να επανέλθει. Όχι, ευχαριστώ. Και πάμε στους, ε, στην ομάδα του EFT. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας, ε, κύριε, ο κύριος Τέρο. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Έχουμε συζητήσει αρκετά ήδη και έχω λάβει τις περισσότερες απαντήσεις που ήθελα. Ίσως λίγες περισσότερες λεπτομέρειες, σας παρακαλώ. Φαίνεται να είναι μια γενική αντίληψη πλέον πως η Ελλάδα θα χρειαστεί ακόμα κάποια μορφή βοήθειας. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση του εύρους της βοήθειας, πόσα δηλαδή, ποιο θα είναι το τρίτο πακέτο, ποιο θα είναι μάλλον ε, το μέγεθος του τρίτου πακέτου bailout και θα, θα γίνει ξανά κούρεμα ή όχι. Και από τον Μπέιλιν τι περιμένετε. Ειλικρινά δεν μπορώ να σας πω και δεν είναι επειδή δεν θέλω να πω, αλλά δεν μπορώ, δεν δύναμε. Γιατί νομίζω πως το ερώτημά σας ρωτά για τη μελλοντική ε, με βοήθεια μετά από αυτό το πρόγραμμα. Εγώ για την ώρα ασχολούμαι με τη συνέχιση αυτού του προγράμματος που ισχύει μέχρι το τέλος του έτους. Και εδώ σε αυτή την περίοδο έχουμε θέματα. Το πρώτο είναι βεβαίως το να πετύχουμε επιτυχώς την ε, τρέχουσα αναθεώρηση. Ελπίζω πως θα έχουμε τα αποτελέσματα το Μάρτιο και θα τα συζητήσουμε στο Eurogroup το Μάρτιο. Και όσον αφορά το ερώτημα το πόσα χρήματα θα χρειαστούν το μέλλον, στο μέλλον δεν μπορώ να πω. Εξαρτάται πάρα πολύ από την ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους που θα κάνουμε αργότερα φέτος. Εξαρτάται πώς θα εξελιχθούν οι δείκτες για την οικονομική ανάπτυξη και θα πρέπει να επανέλθουμε αργότερα. Αλλά το θέμα της βιωσιμότητας του χρέους, ώστε να είμαστε βέβαιοι πως η Ελλάδα μακροπρόθεσμα θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο εθνικό της χρέος, είναι το θέμα κλειδί. Μάλιστα. Και για την Τρόικα, για την Τρόικα τι περιμένετε από την επόμενη της αποστολή. Πάντα πρέπει να προσέχω πολύ για την Τρόικα γιατί νομίζω ότι το γεγονός ότι αυτή η αποστολή έχει κρατήσει τόσο πολύ δείχνει πως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και καταλαβαίνω απόλυτα την δυσκολία της κοινωνικο-οικονομικής και πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα. Και ωστόσο πρέπει να προχωρήσουμε ώστε να ε, μπει σε μια τροχιά βιώσιμη η οικονομία και τα οικονομικά της χώρας. Πρέπει να συνεχιστεί λοιπόν η προσπάθεια. Οι συνεισθητήσεις θα συνεχιστούν τρίτη, Δευτέρα, Κυριακή, Δευτέρα. Πρέπει να υπάρξει ε, πρόοδος πριν να μπορέσει να επανέλθει η Τρόικα στο Eurogroup, γιατί διαφορετικά δεν έχουμε βάση για να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ και τώρα εξ ονόματος του ΕΛΚ, η Καρίν Φόρτμαν Κόλ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, Πρόεδρε του Eurogroup. Ευχαριστώ που βοηθάτε να προχωρήσουν τα πράγματα, να βρεθεί μια λύση για τον νέο μηχανισμό εξυγένσης. Και η Ελλάδα προσπαθεί να πετύχει μια λύση, αλλά πρέπει να πω ότι ο ρυθμός με τον οποίο προχωρά ο τριμερής διάλογος θυμίζει μάλλον σαλιγκάρι. Πρέπει να πάμε πιο γρήγορα. Εσείς βέβαια διπλωματικά αναφερθήκατε στα περιθώρια βελτίωσης, αλλά περιθώρια βελτίωσης δεν βλέπουμε το Κοινοβούλιο θέλει να μην είναι οι χώρες μέλη, αλλά η αρχή του ενιαίου αυτού μηχανισμού να αποφασίζει. Εσείς είσαστε διατεθειμένος ε, να προσπαθήσετε να βρείτε μια λύση από αυτού μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Είναι πολύ σημαντικό για να γίνει αποδεκτή και η διακυβερνητική σας ε, μέθοδος. Δεύτερον, από την αρχή λέμε ότι οι αρχές του μηχανισμού πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν. Πρέπει, ήδη κρατάει πολύ καιρό το χτίσιμο του μηχανισμού αυτού, γιατί πρέπει να υπάρξει διευκόλυνση δανεισμού με τον EFSM. Εσείς βλέπετε ότι μπορεί εκεί να επιτευχθεί μια λύση ή να υπάρξει κοινοτικό ταμείο. Θα προχωρήσετε σε λύση από αυτού. Και μια τελευταία ερώτηση, ξέρω ότι είναι πολλά για πέντε λεφτά. Εσείς δείξατε ηγετικό ρόλο πράγματι όσον αφορά το Eurogroup και για τη, διακυβερνητική, μάλλον για τη διακυβέρνηση. Ε, υπάρχουν το δίπτυχο, το εξάπτυχο κτλ. Εσείς τι θέλετε να πετύχετε τελικά για την μακροοικονομική διακυβέρνηση Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Καταρχήν, όταν λέω ότι υπάρχει χώρος για βελτίωση, δεν είναι μόνο μία διπλωματική έκφραση. Ε, πιστεύω σίγουρα πως μέσα στο πλαίσιο της ε, διαδικασίας λήψης αποφάσεων υπάρχει χώρος για βελτίωση. Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε να σας πω εγώ τι νομίζω προσωπικά, αλλά τι θέλει μάλλον το Eurogroup. Είναι λίγο νωρίς για να σας πω, αλλά έχω καταλάβει ότι πολλές φορές και εξάλλου οι συζητήσεις του ΕΚΟΦΗΝ ήταν δημόσιες και εσείς λέτε να είναι ανοιχτές οι συζητήσεις, όπου είμαι βέβαιος ότι την παρακολουθήσατε και ότι Έγιναν διάφορες προτάσεις από διάφορους υπουργούς για το πώς να βελτιωθούν όλα αυτά. Τώρα πρέπει να δούμε πώς θα δουλέψουμε και πώς θα βρούμε την κατάλληλη στήριξη στο ΕΚΟΦΗΝ και επ' αυτού θα εργαστούμε. Τώρα, σε σχέση με την δανειακή διευκόλυνση και αυτό συζητήθηκε. Και εγώ ως Υπουργός Ολλανδός το ζήτησα, στο, το υπστήριξα στο ΕΚΟΦΗΝ αλλά τώρα ξέρω πως ε, γίνεται συζήτηση για την ε, τμήματοποίηση αυτό σημαίνει πως και οι εθνικές κυβερνήσεις θα είναι υπεύθυνες. Ξέρω το Κοινοβούλιο είναι κατά του να υπάρξει τμήματοποίηση. Θα πρέπει να γίνει και πολύ τεχνική εργασία αλλά μπορεί αυτό τελικά να είναι το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα για την οικονομική διακυβέρνηση, ε, το νόημα των όσων είπατε Δευτέρα είναι ότι βασικά αυτό που έχουμε τώρα, δηλαδή οι ε, αποτελεσματικοί μηχανισμοί που έχουμε τώρα από την πλευρά τη δημοσιονομική θα μπορούσαμε να τους χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους μηχανισμούς και τη μόχλευση που προκύπτει από αυτούς για να προωθήσουμε τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Επίσης ζήτησα συντονισμό ε, σε αυτό το επίπεδο, γιατί τώρα όλοι μας εργαζόμαστε, ας πούμε, για τη μεταρρύθμιση των συντάξεων, αλλά χώρια ο καθένας. Ενώ έχουμε πολλά να μάθουμε και να κερδίσουμε εάν τα κάνουμε αυτά ε, παράλληλα και ταυτόχρονα ε, σε συγκεκριμένο πλαίσιο και χρόνο. Ας πούμε, Ας πούμε, ο τρόπο με τον οποίο αναπτύξαμε την Τραπεζική Ένωση είναι ένα ενδιαφέρον πρότυπο για να το εξετάσουμε και σε άλλου οικονομικού τομείς, όπου η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη θα μπορούσε να ενισχυθεί. Προσπαθώ λοιπόν να είμαι πολύ πρακτικός. Πιστεύω πως τα μέσα που έχουμε μας δίνουν κάποιο εφέ μόχλευσης είναι αποδοτικά για τον προπολογισμό, για τους προϋπολογισμούς, για τα δημοσιονομικά, μήπως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για τις διευθυντικές μεταρρυθμίσεις γιατί πιστεύω πως έχουμε πολλά να κερδίσουμε όσον αφορά την οικονομική μεγέθυνση, η ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, πρέπει εδώ να δω ποιον θα δώσω το λόγο, γιατί ο Κουσόφ δεν είναι εδώ. Επόμενος είναι ο Διόγκο Φιέο. Φέιο, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Κύριε Πρόεδρε, Θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντά σας για την ανάλυση που κάνατε για την λειτουργία των συστημάτων της Τρόικα. Ήταν μια επίγουσα απάντηση που χρειάστηκε να δώσει η Ευρώπη ενώπιον ενός συνόλου συγκυριών που έτρεχαν και θα ήθελα λοιπόν να δω Ποια είναι η γενική σας ανάλυση όσον αφορά τη λειτουργία αυτού της ε, ε, όλης διαδικασίας. Δεύτερον, εάν με βάση την ανησυχία που έχουμε εδώ στο Κοινοβούλιο για τη σειρά ανησυχιών που έχουμε εκφράσει, αν πιστεύετε πως είναι δυνατόν να προχωρήσουμε προς μια λύση που να είναι αυστηρά ευρωπαϊκή, που να μην χρειάζεται για παράδειγμα η επέμβαση, η παρέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το μέλλον. Αυτό ως πρόβλεψη για το μέλλον. Αν προκύψουν δηλαδή ξανά τέτοιες καταστάσεις που ελπίζουμε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπορεί η ευρωπαϊκή απάντηση από εδώ και στο εξή να είναι αποκλειστικά ευρωπαϊκή, που θα δοθεί αποκλειστικά από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ για την Τρόικα. Φυσικά περιμένω την ε, ολοκλήρωση της εκθέσεως του Κοινοβουλίου για την αξιολόγηση της λειτουργίας της Τρόικας και κατάλαβα ότι θα ψηφίσετε γι' αυτό τον Μάρτιο. Η Τρόικα και η όλη προσέγγιση στη διάρκεια της κρίσης ήταν κάτι που επιβλήθηκε από την οξία κρίση τον, ε, που έπληξε τη, τη διακυβέρνηση της κυβερνήσης και το γεγονός ότι οι τράπεζες δεν είχαν πλέον πρόσβαση σε πιστώσεις, αναπτύχθηκαν διάφορα μέσα και το, η Τρόικα έπαιξε βασικό ρόλο πάντοτε υπό την, ε, ε, υπό την πολιτική εποπτεία και την λόγοδοσία στο Eurogroup. Εγώ θα ήμουν ε, πολύ αυστηρός αν τώρα κατηγορούσε κανείς την Τρόικα για τις οικονομικές δυσκολίες των διαφορών χωρών, γιατί αυτές προήλθαν βασικά από οικονομική και πολιτική δυσδιαχείριση, κακοδιαχείριση, πριν να συμβεί η κρίση. Δεύτερον, όποια μέτρα λήφθησαν στη διάρκεια των προγραμμάτων, σχεδιάστηκαν και λήφθησαν αποφάσεις εντός του Eurogroup και όχι από την ίδια την Τρόικα. Φυσικά υπήρξαν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις χώρες και στην Τρόικα στη διάρκεια όλων αυτών και ευτυχώς που έγινε αυτό για να μπορέσουμε πιο συγκεκριμένα να προσαρμόσουμε τα προγράμματα. Αλλά όπως σας είπα πάντοτε αυτό γινόταν υπό την πολιτική καθοδήγηση και έλεγχο του Eurogroup. Και έτσι βλέπω και τη διαδικασία εν γέννη Ευχαρίστω να απαντήσω και σε πιο ειδικευμένε ερωτήσεις. Τώρα όσον αφορά τον μελλοντικό σχεδιασμό, δεν υπάρχει κάποια γενική γνώμη ακόμα στο Eurogroup ότι δηλαδή θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο ε, αποκλειστικά από ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θα μπορούσε να είναι δυνατόν στο μέλλον, αλλά πιστεύω και θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου μάλιστα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην προσπάθεια που κατέβαλε ε, στο να μας βοηθήσει στη διάρκεια της κρίσης. Όχι μόνο με χρήματα αλλά και με εμπειρογνωμοσύνη. Δεν έχω καμιά επίκριση προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τώρα, αν το στο μέλλον θα έχει ακόμα να παίξει κάποιο ρόλο, δεν το γνωρίζω. Θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Δεν υπάρχει κοινή θέση για αυτό το θέμα ακόμη στο Eurogroup. Πρόεδρος, Φαίνεται κάπως να πρέπει να κάνουμε το ζογκλέρ εδώ με τον κατάλογο των ομιλητών και με το ρολόι. Προσπαθούμε πάντα να βελτιώσουμε τα πράγματα. Τώρα, από τους σοσιαλιστές, ένας από τους, εκθε... από τους μας για την Τρόικα. Ευχαριστώ, Σάρων. Κύριος Νόγκ, μου δίνεις ακριβώς την κατάλληλη στιγμή το λόγο. Με την ε, ακρόαση των εκπροσώπων της Τρόικα διαπιστώνουμε ότι τα τελευταία, το τελευταίο διάστημα είχαν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ τους και πολλοί από αυτούς μας είπαν, όπως και εσείς επιβεβαιώνετε τώρα, είπαν στο Eurogroup, μας είπαν ότι λαμβάνονται αποφάσεις στο Eurogroup. Και ως εκ τούτου γι' αυτό κάνουμε τις ερωτήσεις προς εσάς. Λυπούμαστε που δεν ε, δώσατε συνέχεια στο αίτημά μας ε, για ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής ΕΚΟΝ της Υποεπιτροπής για την έρευνα για την Τρόικα, για τον ρόλο τη Τρόικα. Αλλά μια και είστε εδώ θα σα κάνω τώρα τι ερωτήσει. Πρώτα λοιπόν και από τα όσα έχουμε δει και από τα ταξίδια μα ε, στι χώρε, θα ήθελα να σα ρωτήσω τα εξή για την Κύπρο. Ποιο από το Eurogroup πρότεινε την φορολόγηση των μικροκαταθετών κάτω από τι 100.000 ευρώ μέτρο το οποίο ευτυχώ απερίφθη από το Κυπριακό Κοινοβούλιο παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Συνθήκη, αλλά θέλω να ξέρω ποιος έκανε την πρόταση στο Eurogroup. Δεύτερον, η Ιρλανδία. Μας εξηγήσατε ότι τα πάει καλά η Ιρλανδία. Πλην όμως, όταν πήγαμε εμείς στην Ιρλανδία και συναντηθήκαμε με τον κύριο Νούναν, Υπουργό των Οικονομικών, και μάλιστα ο κύριος Νούναν τώρα κάνει μια πρόταση δημοσία για τη μεταφορά. Σας παρακαλώ ο κύριος Νούναν κάνει μια πρόταση δημοσία για τη μεταφορά μέρους των, του Ιρλανδικού χρέους ε, στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για να αντιμετωπίσει ακριβώς την ε, τραπεζική κρίση. Η δε κυρία Μπόλς, δίπλα σας προτείνει το τμήμα των δημοσίων αποφάσεων που αφορούν την ε, επιστροφή του χρέους να βγει από τον υπολογισμό του δημοσίου χρέους. Έτσι λοιπόν, ώστε, του δημοσίου ελλείμματος. Έτσι λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, τι συνομιλίε έχετε με την Ιρλανδική κυβέρνηση, τι λύσεις προτείνετε για την Ιρλανδία ώστε να περιοριστεί αυτό το τραπεζικό χρέος που επιβαρύνει τόσο σημαντικά τον φορολογούμενο, δεδομένου ότι την εποχή που αποφασίστηκε δεν υπήρχαν οι σχετικοί μηχανισμοί διάσωσης. Τελευταία ερώτηση για την Ελλάδα, διότι δεν απαντήσατε στους συναδέλφους και κυρίως τον κύριο Κλούτε ναι, όντως η Ελλάδα θα έχει πρωτογενές πλεόνασμα, κάνει τις απαραίτητες προσπάθειες για να εξασφαλίσει το πρωτογενές πλεόνασμα και φέτος θα ξαναβρει το δρόμο της ανάπτυξης. Αλλά η κυρία Λαγκάρτ δηλώνει στο Financial Times, και αυτή είναι η θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ότι μακροπρόθεσμα το χρέος της Ελλάδας, εάν μείνει άνω του 120% του ΑΕΠ, δεν είναι βιώσιμο. Τώρα έχει φτάσει στα 175%. Η θέση του Δούνου του εξ αρχής ήταν να ζητήσει ανάταξη του ελληνικού χρέους. Ερωτώ λοιπόν, επιβεβαιώνεται ότι αυτή τη στιγμή προκύπτει διάλογο στο Eurogroup και ο κύριος Τουρνάρας μας επιβεβαίωσε ότι γινόντουσαν συνομιλίες προκειμένου να απλωθεί χρονικά το ε, χρέος της Ελλάδας και να μειωθεί το επιτόκιο εφόσον εξασφαλίσει πρωτογενές πλεόνασμα η χώρα. Μας επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι ξεκινάει αυτός ο διάλογος στη Eurogroup. Και σταματάω εδώ, δεν θα έχετε το χρόνο να απαντήσετε. Απάντηση. Εντάξει, πολύ. Ήταν πολύ εκτεταμένες οι απαντήσεις σας και δεν θα έχω χρόνο. Επαρκεί. Καταρχάς, ε, κάνατε την παρατήρηση ότι δεν ήρθα να μιλήσω για την Τρόικα στο Κοινοβούλιο. Να σας πω, η ερώτηση για την Κύπρο μου υπευλήθη την προηγούμενη φορά ή την προ-προηγούμενη που ήρθα να μιλήσω στην Επιτροπή σας. Ακριβώς την ίδια ερώτηση. Ποιος πρότεινε να φορολογηθούν οι μικροκαταθέσεις. Ο κύριος Έικχαουτ ή κάποιος άλλος από την Επιτροπή σας είχε καταθέσει την ερώτηση, θα σας δώσω και την ίδια απάντηση που είχα δώσει και τότε, η οποία είναι ότι δεν έχω την δυνατότητα, δεν δικαιούμαι να αποκαλύψω ποιος πρότεινε τι στην συζήτηση του Eurogroup. Όπως είπαμε, προέκυψε μια απόφαση, μια πρόταση καλύτερα από την πρώτη αυτή συνεδρία του Eurogroup, δεν επέτυχε και πολύ γρήγορα ελήφθη μια άλλη απόφαση επίσης πολύ σκληρή για την Κύπρο και τις τράπεζές της. Αλλά βέβαια το σημαντικό είναι εγώ να στηρίξω το αποτέλεσμα και να μην επισέλθω στην αποκάλυψη του ποιος είπε τι. Αυτό όμως αναπάτησε το έχω δώσει εδώ και μήνες. Ιρλανδία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχει σημαντικά επιβαρυνθεί ο φορολογούμενος, ο πολίτης από το χρέος του τραπεζικού τομέα στην Ιρλανδία, εάν υπήρχαν τα κατάλληλα εργαλεία διάσωσης ε, την εποχή εκείνη, θα ήταν η κατάσταση διαφορετική για τους Ιρλανδούς πολίτες. Η αναδρομική χρήση της άμεσης ανακεφαλοποίησης από το με μηχανισμό σταθεροποίησης είναι κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε. Συζητούμε ούτως ή άλλως ήδη. Είναι κάτι το οποίο έχει μείνει ανοιχτό από την απόφαση του Ιουνίου η δυνατότητα ανακεφαλοποίησης από τον μηχανισμό σταθεροποίησης. Υπάρχουν κάποιες τάσεις να συζητηθεί το κατά πόσο είναι επιθυμητό αυτό, χωρίς να μπορώ να προκαθορίσω ή να προδικάσω την απόφαση. Πάντως υπάρχουν οι δυνατότητες από την απόφαση του Ιουνίου να καλυφθεί η ανακεφαλοποίηση από τον μηχανισμό σταθεροποίησης για την Ελλάδα το αν είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα το χρέος ή όχι. Όταν αποφασίσαμε το πρόγραμμα προσαρμογής το 2012, το Δεκέμβριο, έκαναμε τους υπολογισμούς της βιωσιμότητας του χρέους μαζί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με στόχευση το 124% το 2022. Αυτό είχε υπόψη και το δούνου του ως βιώσιμο χρέος. Βραχυπρόθεσμα μπορεί να είναι υψηλότερο του 124% επί του ΑΕΠ μεν, αλλά μακροπρόθεσμα έως το 2022 θα μειωθεί στο 124%. Βέβαια στο τέλος του έτους θα ξαναγίνει ο υπολογισμός, θα ξαναυπολογιστεί η βιωσιμότητα του χρέους, θα δούμε πού βρισκόμαστε και αν οι συνθήκες στις οποίες συμφωνήσαμε το Δεκέμβριο του 2012 δεν ισχύουν πλέον, θα πρέπει να συζητήσουμε τους όρους αυτούς και να προσφέρουμε περαιτέρω υποστήριξη στην Ελλάδα να είμαστε διατεθειμένοι να υποστηρίξουμε περαιτέρω την Ελλάδα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σα βεβαιώσω ότι ο στόχο αυτό, τον οποίο στα τέλη του 2012 είχαμε συμφωνήσει με το Διεθνέ Σωματικό Ταμείο, τηρείται ακόμη εντό των προθεσμιών ή όχι. Θα πρέπει να επανέλθουμε στα τέλη του τρέχοντος έτος για να συζητήσουμε την βιωσιμότητα. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο και τώρα περνάμε στου άλλου συνεισηγητέ για την Τρόικα, για, στον άλλο συνεισηγητή για την Τρόικα, Ότμαρ Κάρα, εάν θε να πει κάτι. Κύριε Ντάιζεμπλουμ, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο πτυχές. Αφενός μεν αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πρόβλημα πάντα όταν στην απάντησή σας επικαλείστε μηχανισμούς και θεσμούς που δεν ρυθμίζονται από το κοινοτικό δίκαιο. Δεν θα ήταν λοιπόν πολύ πιο απλό το να είστε σε θέση να μας πείτε ότι κάθε διακυβερνητικό όργανο και δραστηριότητα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά έργα και τους στόχους παραμένουν σε εθελοντική βάση μέχρι τροποποίησης της συνθήκης. Γιατί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας μπορεί να εδρεωθεί στο κοινοτικό δίκαιο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Οι κανόνες του το επιτρέπουν. Εμείς λοιπόν προτείνουμε να ενημερωθεί η Τρόικα, να συμπληρωθεί η Τρόικα με ένα μηχανισμό καινούριο που θα την εδραιώνει στο ευρωπαϊκό ε, ρυθμιστικό πλαίσιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη. Οπότε δεν έχουμε ούτε για λογοδοσία, ούτε για διαφάνεια, ούτε για νομιμότητα κανένα πρόβλημα. Ποια είναι η θέση σας λοιπόν σε αυτό. Και επίσης αναφερθήκατε στην ανεργία. Συζητάτε πάλι το θέμα των χρηματοπιστωτικών φόρων στο ΕΚΟΦΗΝ, ενώ από τον Ιούλιο έχει υποστηρίξει την πρόταση αυτή το Κοινοβούλιο, 57 δισεκατομμύρια ευρώ χάνονται βάσει μελετών επειδή δεν επιβλήθη ο, ε, χρηματοπιστωτικό, ο φόρος στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Λέτε ότι θέλετε να, καταπολεμήσετε την ανεργία, θέλετε την, ε, την ανάπτυξη, θέλετε την απασχόληση. Πώς λοιπόν μπορεί, αυτε, μπορείτε αυτές τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να τις υλοποιήσετε και πότε. Απάντηση. Θέλετε δηλαδή όλα τα διακυβερνητικά ε, έργα, εγχειρήματα κτλ. προς το παρόν να γίνουν σε εκούσια βάση, όπως λέτε, με εδραίωση στην κοινοτική μέθοδο. Δεν ξέρω αν είναι δυνατόν αυτό. Ως πρόεδρος του Eurogroup εγώ στηρίζομαι στους κανόνες και τις ρυθμίσεις που έχουν διακυβερνητική βάση και λογοδοτώ ως υπουργό, όπως και οι άλλοι, στα Εθνικά Κοινοβούλια. Δύο φορές το χρόνο τουλάχιστον έρχομαι στην Επιτροπή σας το γνωρίζετε αυτό, αλλά αυτό βέβαια είναι κάτι άλλο από την κοινοτική μέθοδο που επικαλείστε. Επομένω, βασικά πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα όπω το έχουμε σχεδιάσει. Ναι, βεβαίω είναι υβριδική αυτή η ένωση και μακροπρόθεσμα ασφαλώ θα έχει κάποια εξέλιξη, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά ω πρόεδρος του Eurogroup δεν είμαι σε θέση να προχωρήσω εγώ με δική μου πρωτοβουλία σε διαφορετική μέθοδο, δεν θα ήταν σωστό κάτι τέτοιο. Για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών υπάρχει μια ομάδα ενισχυμένης συνεργασίας 11 κρατών μελών που προσπαθούν τώρα να βρουν μεταξύ τους μία λύση για τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο έχουν προχωρήσει, διότι εγώ δεν συμμετέχω στην ομάδα αυτή ως Ολλανδός υπουργό των Οικονομικών, ούτε βέβαια ως πρόεδρος του Eurogroup θα μπορούσα να συμμετάσχω. Όταν λάβουν απόφαση τότε θα μπει στην ημερήσια διάταξη του ECOFIN, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό της οριμότητας της συζήτησης, ώστε να μπει στην ημερήσια διάταξη του Eurogroup. Αυτό γνωρίζω. Ξέρω ότι δεν σας ικανοποιεί η απάντησή μου, αλλά εγώ δεν εμπλέκομαι ούτε ως υπουργό της Ολλανδίας, ούτε ως πρόεδρος του Eurogroup στην ομάδα αυτή ενισχυμένη συνεργασία και έτσι δεν γνωρίζω τι συζητούν. Για το ποσό το οποίο αναφερθήκατε, δεν ξέρω ακριβώ να το επιβεβαιώσω, ή μιλάτε πάντω για δισεκατομμύρια που χάνονται λόγω τη μη υλοποίηση του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Μα όχι, δεν είναι χαμένα τα λεφτά αυτά, πάνε αλλού στην οικονομία, κάπου αλλού αξιοποιούνται. Από εκεί και πέρα, εάν θέλει πολιτικό, η πολιτική να τα φορολογήσει στην πηγή που λέγεται χρηματοπιστωτική συναλλαγή, έχει καλώ. Ιδάλω όμω μπορεί να τα φορολογήσει και αλλού. Πάντω δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο προ το παρόν, γιατί δεν ανήκω, δεν συμμετέχω σε αυτή την ομάδα ενισχυμένη συνεργασία. Επόμενο, Άντωνη Πρεσέντα, εκ μέρου των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ. Κάτι γενικό πρώτα και μετά πιο συγκεκριμένα. Το γενικό είναι το εξή. Έχουμε την τρίμηνη έκθεση της Επιτροπής και του ΩΣΑ της Επιτροπής λέει ότι προβλέπεται τα επόμενα 10 χρόνια μια ανάπτυξη μικρότερη από εκείνη των ετών που είχαμε πριν από την κρίση. Η Ευρώπη δηλαδή είχε πάει χειρότερα από ό,τι οι υπόλοιποι στον κόσμο. Και ότι θα είμαστε στο 1 τρίτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ ο ΣΑ λέει ότι οι προσαρμογές στους μισθούς επηρεάζουν τις τιμές. Τι βλέπουμε λοιπόν, βλέπουμε την ανεργία, τις αλλαγές στους μισθούς, τις μειώσεις, αλλά δεν βλέπουμε μείωση στις τιμές. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, στις Ηνωμένε Πολιτείε η κυρία Γέλεν του ΦΕΔ πήγε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και εκεί μίλησε για τις τιμές και τη σχέση με την απασχόληση. Το θέμα όμως αυτό τελικά δεν βοηθάει τους ανθρώπους. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι είμαστε σε ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση και ότι δεν μπορεί να συνεχίζουμε έτσι. Είμαστε σε μια βαθιά κρίση και ότι τελικά χωρίς ισορροπία επομιζόμαστε τα βάρη. Για το θέμα της Ελλάδας τώρα πιο συγκεκριμένα. Η Ελλάδα εντάξει έχει διάφορες ασθένειες, υποθερμία κλπ. Αλλά όποιο έχει υποθερμία δεν το βάζουμε στο ψυγείο. Συνεπώς νομίζω ότι και εσείς έχετε κάποια ευθύνη απέναντι στην Ελλάδα. Πολλά λέμε, αλλά εσείς θα αναλάβετε τις δικές σας ευθύνες απέναντι στην Ελλάδα. Τρίτον, τι θα γίνει μετά τα προγράμματα προσαρμογής. Η Ισπανία, ολοκλήρωσε το μνημόνιο, η Ιρλανδία, εντάξει, τα τηρήσαμε. Τώρα, τι θα γίνει για να προστατευτούμε απέναντι στο μέλλον. Και ο μηχανισμός σταθερότητας, εσύ είπατε ότι μπορούμε να σας ρωτήσουμε για αυτό το θέμα, μα η καλύτερη ερώτηση είναι εξή. Είναι μηχανισμός για τη σταθεροποίηση τη Ευρωζώνης εμείς θα φτιάξουμε ένα φύλλο πορείας ώστε να γίνει αυτό σε κοινοτικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Για την οικονομική ανάπτυξη. Νομίζω ότι έχετε δίκιο. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτό το χαμηλό διορθωτικό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης για την Ευρώπη. Γιατί, Γιατί δεν θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε την ανεργία με το ρυθμό που θέλουμε να το κάνουμε και δεν θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα δημοσίου χρέους με το ρυθμό που θέλουμε να το κάνουμε. Συνεπώς, πρέπει να έχουμε την φιλοδεξία να πετύχουμε μεγαλύτερα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης. Και γι' αυτό και είπα ότι στο Eurogroup υπογραμμίζουμε ιδιαίτερα το θέμα της διαχείρισης της κρίσης, προγράμματα κλπ. Δημοσιονομικά οι προπολογισμοί δηλαδή να είναι εντάξει, αλλά υπογραμμίζουμε επίσης ότι σιγά σιγά πρέπει να ασχοληθούμε και με τους στόχους της οικονομικής ανάπτυξης. Και σας είπα υπάρχει δυναμικό. Δεν νομίζω ότι πρέπει να δεχτούμε αυτά τα χαμηλά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης, γιατί υπάρχουν δυνατότητες, αρκεί βέβαια να ε, υπάρξει μεταρρύθμιση στην στρατηγική μας. Για την κάθε χώρα ισχύει κάτι διαφορετικό. Η κάθε χώρα πρέπει να κάνει κάτι διαφορετικό για να αντιμετωπίσει τις διευθυντικές ανισορροπίες. Εσείς είπατε ότι σε πολλές χώρες, ιδιαίτερα στη Νότια Ευρώπη, μειώθηκαν οι μισθοί, το κόστος εργασίας μειώθηκε, όχι όμως και οι τιμές. Αυτό τι δείχνει. Δείχνει ότι οι αγορές ανατομέα, αγορές προϊόντων δεν λειτουργούν. Γιατί αν μειώσετε το επίπεδο τιμής παραγωγής, ε, προφανώς πρέπει να μειωθούν και τιμές. Δεν έγινε όμως αυτό, άρα οι αγορές δεν λειτουργούν. Υπάρχει συνεπώς μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και πάρα πολύ συγκεκριμένοι στην ανάλυση μας ανά χώρα για να δούμε πού υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και τι μπορούμε να κάνουμε. Μέχρι τώρα αυτό έχει μείνει στις εθνικές κυβερνήσεις και μόνο αν υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης ολόκληρη την ΟΝΕ ναι, και στις άλλες χώρες, τότε μόνο παρεμβαίνουμε. Αλλά κατά τη γνώμη μου και τη Δευτέρα είπα ότι αυτή είναι μια αμυντική προσέγγιση. Δηλαδή μόνο αν υπάρξει κάτι αρνητικό παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει τι πρέπει να κάνετε για να διαρθρώσετε τις οικονομίες σας. Ενώ πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί εντό αγωγικών και να μιλήσουμε για όλα τα θέματα που είναι στην ημερήσια διάταξη για όλες τις χώρες, είτε πρόκειται για τα συνταξιδιωτικά και το, την ηλικία συνταξιδότηση, είτε πρόκειται για την αγορά προϊόντων. Εκεί πρέπει να υπάρχει συνεργασία για να πετύχουμε αυτό το υψηλότερο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν επιμένω υπάρχει μεγάλο περιθώριο και δυναμικό για ανάπτυξη και δεν πρέπει να το παραβλέπουμε αυτό. Δεν έχω άλλο χρόνο για να απαντήσω σε άλλες δύο ερωτήσεις, λυπάμαι. Πρόεδρος, ναι, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι πιέζει ο χρόνος. Συνεχίζουμε. Ίσως βρείτε χρόνο να απαντήσετε και σε αυτές τις ερωτήσεις και για την Ελλάδα και λοιπά. Για το ΕΛΚ, Τόφμαν, Χέρμπαρτ, είδα που είσαι. Α, εκεί, ναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ερώτησή μου αφορά τις ανισορροπίες στο χώρο του ευρώ. Νομίζω ότι και τα διαφορετικά επιτόκια που προσφέρονται από τις τράπεζες για τις ιδιωτικέ μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις είναι ένα πρόβλημα. Οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορεί να βρουν έναν τρόπο χρηματοδότηση στο διεθνές, στη διεθνή αγορά, αλλά οι ιδιωτικές μικρές και μεσές επιχειρήσεις ε, εξαρτώνται από την εθνική αγορά χρήματος, το ΣΥΠΗΝ. Εγώ δεν είμαι σε θέση ε, στην Ιταλία όπου βρίσκομαι ως επιχείρηση να στραφώ ε, από την Ιταλία στην οποία βρίσκομαι ως επιχείρηση να στραφώ σε μια Αυστριακή που βρίσκεται 50 χιλιόμετρα μακριά μένα αλλά από την άλλη μεριά των εθνικών συνόρων για να εξασφαλίσω χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε κάποιους τρόπους να εξασφαλίσουμε καλύτερε ισορροπίες σε αυτό και επίσης ε, τα επιτόκια αυτά βλέπουμε να έχουν να παρουσιάζουν ψαλίδα μεγάλη τους τελευταίους μήνες που δεν κλείνει. Μια ευρωπαϊκή αγορά χρήματος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, χρειάζεται όμως να την εξασφαλίσουμε, να μπορούμε να εξασφαλίσουμε την χορήγηση ε, δανείων πέραν των συνόρων και αυτό βέβαια προϋποθέτει την ασφάλιση του δανείου, δηλαδή την εγγύηση. Και αυτό χρειάζεται ένα νομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ τα αναγνωρίζω αυτό που λέτε, ότι η ερμηνεία συνεχίζεται. Δεν τα έχω δει τα δεδομένα, αλλά το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς πιστώσεων μπορεί να είναι το αποτέλεσμα τελικά της δημιουργίας της Τραπεζικής Ένωσης. Βέβαια υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία εξηγούν τις διαφορές στα επιτόκια, οικονομικό ρίσκο ή το ποσό πιστώσεων που μπορεί να προσφέρει ένας τραπεζικός τομέας, ή τράπεζες. Έχει να κάνει λοιπόν με την πραγματική οικονομία αντικατοπτρίζει τον κίνδυνο στις αγορές ή έχει να κάνει και με την, ε, τον κατακαιρματισμό του δημοσιονομικού τομέα στην Ευρώπη. Κατακαιρματισμό. Υπάρχει, το είδαμε αυτό και με την Τραπεζική Ένωση προσπαθούμε να φτιάξουμε. Ο λόγο που προσπαθούμε να το φτιάξουμε αυτό, την Τραπεζική Ένωση, είναι ότι θέλουμε να έχουμε ένα σταθερό αλλά και ενιαίο δημοσιονομικό τομέα στην Ευρώπη και η γη, βέβαια. Καλώς, ευχαριστώ. Θέλετε να επανέλθετε. Πολύ σύντομα. Α, βεβαίως. Αντιλαμβάνομαι ότι οι διαφορέ στα επιτόκια μπορεί να εξηγούνται ή να έχουν σχέση με μια οικονομική κατάσταση σε μια χώρα. Αλλά σα έδωσα το συγκεκριμένο παράδειγμα. Σε λίγα χιλιόμετρα απόσταση από τα σύνορα, μια μικρομεσαία επιχείρηση θα έπρεπε να μπορεί να πάει σε μια γειτονική τράπεζα του γειτονικού κράτους όμως, μερικά χιλιόμετρα μακριά όπως λέω, για να, λέω, για να ζητήσει τη χρηματοδότηση. Εάν μπορούσε να υπάρχει σχετική ε, εξασφάλιση ε, ε, για την τράπεζα. Όταν έχουμε λοιπόν μια κοινή αγορά πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για τις τράπεζες να δράσουν με πιο ανταγωνιστικό τρόπο μέσα στο τραπεζικό σύστημα. Ναι, έχετε δίκιο. Τμήμα της Τραπεζικής Ένωσης έχει να κάνει και με ένα ενιαίο κανονισμό, μια ενιαία ρύθμιση τραπεζική. Θα πάρει όμως χρόνο. Προς το παρόν έχουμε τις, νομ... νομοθεσίες των χωρών μελών. Αλλά προοδευτικά προχωράμε προς μια τέτοια ενιαία ρύθμιση ώστε να παληθούν οι διασυνοριακές διαφορές που υπάρχουν σήμερα. Αυτό, τίποτα άλλο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Έχουμε καθυστερήσει, τέλο πάντων δεν ξαναβάλα το ρολόι. Τώρα από τους σοσιαλιστές, Λεωνάρντο Ντομίνιτσι. Στα αγγλικά, για να τα πω πιο γρήγορα, λέει ο μιλτής. Χρειάζονται πολλές προϋποθέσεις προκειμένου να αντιληφθούμε την ανάκαμψη στην Ευρώπη. Ένα από τα στοιχεία αυτά έχει να κάνει με την εξισορρόπηση των οικονομιών στην Ευρωζώνη. Πιστεύετε ότι χρειαζόμαστε σημαντική πτώση των μεγάλων νομισματικών πλεονασμάτων που υπάρχουν σε βόρειες χώρες, κατοχώρες και Γερμανία για παράδειγμα. Και συμφωνείτε με αυτή την άποψη. Τι είδου μέσα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Ναι, βλέπω περιθώριο για να βελτιωθεί η ζήτηση στην Ευρώπη εσωτερική ζήτηση από διάφορες χώρες. Και γίνεται, αν δείτε τους μισθούς στη Γερμανία, οι οποίοι αυξάνονται τα τελευταία χρόνια. Το ίδιο θα γίνει και στις κάτω χώρες, κατά πάσα πιθανότητα, τουλάχιστον σε κάποιους τομείς, όταν αρχίσει η οικονομική ανάκαμψη. Ξέρετε, η χώρα μου δύσκολα και αργά βγαίνει από την κρίση. Και γι' αυτό οι μισθοί παρέμειναν με μηδενική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Η ζήτηση πιστεύω ότι θα επιστρέψει πιο δυνατή σε ολόκληρη την Ευρώπη από τις βόρειες χώρες. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να κοιτάμε την Ευρώπη σαν ε, ένα παιχνίδι που λέει ότι συγκινούν το δοχείο, ότι ανάλογα με το τι γίνεται στο νότο θα γίνεται και στο βορρά. Η Γερμανία κάνει χρήμα για όλους μας στην Ασία. Και ελπίζω ότι θα συνεχίσουν να το κάνουν. Επιχειρήσεις από ολόκληρη την Ευρώπη δουλεύουν για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Κατασκευάζουν αυτοχήματα, αυτοκίνητα ή ανταλλακτικά στην Ασία. Οπότε, ναι, παρακαλώ να συνεχίσει αυτό η κάθε χώρα εφόσον μπορεί να εξάγει όπου υπάρχουν ευκαιρίες και δυνατότητες για μας, ναι, είναι καλό αυτό. Ναι, αλλά μια ισχυρή Ευρώπη θέλουμε. Ναι, διπλωματικά απαντάτε τώρα. Το θέμα είναι αν θα υπάρξει υποτίμηση όχι του ευρώ, ε. Τελευταία ερώτηση. Από την Άλντε, ο κύριος Θόδωρος Κελάκης. Παρακαλώ. Thank you, Chair. I will uh, speak in Greece. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, θα μιλήσω αγγλικά. Ελληνικά. Ε, αγαπητέ Πρόεδρε, για την Ελλάδα και με εντυπωσιάσατε. Πρέπει να ζούμε εμείς λίγο κάπως σε άλλη χώρα, γιατί στη δική μας χώρα ο ιδιωτικός τομέας καταστρέφεται από την υπερφορολόγηση και τα ακριβά, πανάκριβα επιτόκια, την ώρα που η ευρωπαϊκή πλευρά συνεχίζει να χρηματοδοτεί κατανοητικές δαπάνες δημοσίου. Πολύ σύντομα κάποια στοιχεία. Έχουμε σήμερα στην Ελλάδα 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενους που δεν πληρώνουν κανονικά τις οφειλές στην εφορία. Ένα εκατομμύριο νοικοκυριά που δεν πληρώνουν κανονικά τις οφειλές τους για ηλεκτρικό ρεύμα. Οι μισοί επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενοι δεν πληρώνουν κανονικά τις εισφορές τους στα ασφαλιστικά ταμεία. Χρωστούν 8 δισεκατομμύρια. 2 εκατομμύρια δάνεια είναι σε καθυστέρηση και πάνω από 500.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα μένουν απλήρωτοι με καθυστερούμενες οφειλές από τις επιχειρήσεις. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς μπορεί ένας συντετριμένος ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα να καταφέρει να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Οι εξαγωγές του 2013 έμειναν στάσιμες παρά το γεγονό ότι όλοι προέβλεπαν ότι θα αυξηθούν και οι μισθοί έχουν πέσει. Πώς θα υπάρξει ανάκαμψη χωρίς εξαγωγές και τέλος γιατί αποδέχτηκε η ευρωπαϊκή πλευρά να μειωθεί φέτος το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην Ελλάδα για να αυξηθεί το πρωτογενές πλεόνασμα που θα μοιραστεί προεκλογικά πρώτων ευρωεκλογών ως, προ, ως ε, παροχές προεκλογικές. I think, um... Νομίζω ότι πολλά από αυτά που αναφέρατε δείχνουν ακριβώς τα θεμελιώδη προβλήματα που υπάρχουν στη λειτουργία του ελληνικού δημοσίου τομέα αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Είναι αδύνατο να έχουμε μια υγιή οικονομία και υγιή δημοσιονομικά αν δεν έχουμε και μια οικονομία και φορολογικό σύστημα που να είναι δίκαιο και στο οποίο όλοι να συνεισφέρουν. Είναι αδύνατον να έχουμε έναν ιδιωτικό τομέα και μια οικονομία που να λειτουργεί αν δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς τους οι πολίτες. Είναι βασικά ζητήματα αυτά. Και υπάρχει με στο πρόγραμμα η αντιμετώπιση του φορολογικού, η αντιμετώπιση των χρεών των πολιτών προς το κράτος. Αλλά έχει να κάνει εδώ και το θέμα της εμπιστοσύνης να συνεισφέρουν οι άνθρωποι σε ένα φορολογικό σύστημα στο οποίο να έχουν εμπιστοσύνη. Είναι θεσμικά ζητήματα αυτά λοιπόν, τα οποία όντω πρέπει να αντιμετωπιστούν. Είναι μέρος του προγράμματος και είναι στοιχειώδη. Αν δεν βελτιωθεί αυτό, και νομίζω ότι βελτιώνεται το φορολογικό σύστημα, για παράδειγμα, πιστεύω ότι έχει γίνει πολλή δουλειά από αυτού για να βελτιωθεί, για να λειτουργεί Όσο δεν γίνεται, εμποδίζει βέβαια την οικονομική ανάπτυξη. Για τους ιδιωτικούς επενδυτές είναι πολύ βασικό. Αν θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση στην Ελλάδα πρέπει να ξέρουν μέσα σε τι φορολογικό σύστημα λειτουργούν και ότι οι λογαριασμοί θα πληρώνονται και από την κυβέρνηση και από τις άλλες επιχειρήσεις. Επανέρχομαι. Δεν έχουν λεφτά για να πληρώσουν το, το ναι. φόρο. Δεν είναι ότι φοροδιαφεύγουν. Δεν έχουν τα χρήματα. Και η πραγματική ερώτηση πίσω από αυτό είναι γιατί δεν, δεν αυξάνονται οι εξαγωγές. Πώς το εξηγείτε αυτό. Πώς μπορείτε να προβλέψετε ανάπτυξη όταν δεν, δεν αυξάνονται οι εξαγωγές. Νομίζω ότι η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας από τις πρόσφατες μελέτες φαίνεται να ε, βελτιώνεται και να επανέρχεται στην ανάπτυξη η χώρα. Θα ήμουν πολύ πιο αισιόδοξο από εσάς. Αλλά το θέμα του φόρου και της φοροδιαφυγής είναι υπαρκτό. Εσύ μπορείτε να, να λέτε ότι δεν μπορούν να πληρώσουν το φόρο τους οι πολίτες. Σε ένα βαθμό μπορεί να ισχύει για πολλούς ε, πολίτες της Ελλάδας. Αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο τμήμα των πολιτών που απλώς δεν πληρώνουν φόρους ή δεν τους πληρώνουν στον απαιτούμενο βαθμό. Και αυτό είναι ένα ζήτημα κρίσιμο για κάθε κοινωνία, για κάθε οικονομία. Προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει κατά τρόπο σωστό πρέπει να έχει και σωστό φορολογικό σύστημα. Γι' αυτό υποστηρίζουμε την Ελλάδα στις προσπάθειές της για να ενισχύσει το σύστημα της φορολογίας. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος, και ευχαριστώ που ήρθατε για αυτόν τον οικονομικό διάλογο. Θα συνεχίσουμε εμεί τώρα με τις ψηφοφορίες μας. Σε λίγα λεπτά θα ετοιμαστούμε, θα ετοιμάσουμε τους καταλόγους των ψηφοφοριών και όλα αυτά. Θα σας αφήσω το περιθώριο λοιπόν αυτό, όσον αποχαιρετήσω τον κύριο Ντάισιμπλουμ. If members could take their seats, then we can do a test. Παρακαλώ, καθίστε για να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. I've, I've, I've opened the vote, so can we check cards are working? Press the happy buttons, please. Um, anybody without a card? Παρακαλώ, όσοι δεν έχετε κάρτες, να μου ειδοποιήσετε, να ξέρω να μετράω. is So we've got 35 plugged in, 34 have pressed their buttons. I'm still waiting. Oh, I can see some abstaining as to whether they're happy or not. Λοιπόν, παρακαλώ να μου δείχνετε αν συμφωνείτε ή όχι. Ψηκάνουμε τη δοκιμαστική ψηφοφορία, ωραία. Λοιπόν, όλα λειτουργούν τα μηχανήματα, πολύ ωραία, για να ξεκινήσουμε με τις ε, ψηφοφορίες μας. Πρώτη είναι η έκθεση του Διόγκο Φέιο. Και η πρώτη τροπολογία είναι η 215. επί αρκατά αποχές απορρίπτεται. 23. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 216 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 217 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 218 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική α υπέρ... Α, με συγχωρείτε. Πρώτο τμήμα, πρώτο τμήμα. Ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε τώρα στην συμβιβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική γ. σι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ε, τροπολογία 283 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 289 υπέρ κατά τι έγινε παιδιά δεν να παρακολουθείτε να πάω λίγο πιο αργά μάλιστα 289. Υπέρ ποιοι είναι, κατά ποιοι είναι. Λυπόμαι, αλλά οι σοσιαλιστές λένε πως είναι υπέρ, αλλά... Λοιπόν, ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο, γιατί μέχρι να πω το κατά, είσαστε υπέρ και γίνεται λίγο μπέρδεμα. The plot, the Και δεν κατάλαβα που είμαστε, ούτε έχω καταλάβει τι παίζει. Λοιπόν, Λοιπόν, ωραία. Α, ναι, τελικά υπέρ ήσασταν. Μπράβο. Πάμε τώρα στην συμβιβαστική ε. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 292 με προφορική Υπέρ αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω πως απορρίπτεται, αλλά θα το ελέγξουμε. 50. One more to vote if you're voting. Uh, no, I'm wrong. That was carried. Άχι, λάθος έκανα, εγκρίθηκε. Ευτυχώς που ελέγξαμε. 295 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 296 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 297 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 298 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 299 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 300 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Α, για να το ελέγξουμε. One more to vote. voting. I'm closing the vote. Ένας ακόμα πρέπει να ψηφίσει. Ωραία, πέρας ψηφοφορίας 22 προς 15 εγκρίνεται. 301 υπέρ κατά αποχές. Δεν είδα τους σοσιαλιστές καν να ψηφίζουν. Τι ψηφίζετε, ας ελέγξουμε. Είναι δύσκολο αν δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Λοιπόν, 301, έλεγχος. Voted, votes closed. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 302 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 303 υπέρ. Ε, κατά. Αποχές. Τα μπέρδεψα. Έλεγχος ηλεκτρονικός. We're checking 303. Έλεγχος για την 303. Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 304 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 305 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 306 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα έχουμε τη συμβιβαστική G. Ναι, Διόγκο. Θέλω μόνο να τονίσω ότι σε σχέση με την προφορική τροπολογία η ομάδα του ΕΛΚΑ θα ψηφίσει υπέρ. Απλώς θέλω να δώσω αυτή την υπόδειξη για να μην, υπάρξουν σύγχυση, να μην υπάρξει σύγχυση. Για την προφορική λοιπόν το ΕΛΚ θα ψηφίσει υπέρ. Thank you very much. I'll uh, Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, συμβιβαστική G με την προφορική τροπολογία πρώτα λοιπόν. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται με την προφορική. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην τροπολογία 313 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. 1919, uh, so that 19-19 Καταπίπτει. Λυπούμε. Α, μπορεί και να μην πρέπει να λυπηθώ. 314. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 315 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 316 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 318 υπέρ κατά να ελέγξουμε την 318 ηλεκτρονικά παρακαλώ Ωραία, τέλος της ψηφοφορίας 19-19 καταπίπτει. 319 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τζόρι 8 έχει καταπέσει, 320 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 53 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 321 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Y ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 328. 328 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 329 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε 429. Three more to vote, two more to vote, two more buttons not pressed yet. Δύο ακόμη ψηφίστε παρακαλώ. 18-18 καταπίπτει. Uh, okay. Who knows what those two unpressed buttons might have done. Uh, 59 in favour. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 330 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 331 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος του 331. One more button if you're pressing. Okay, I'm closing the vote. And that... Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 332 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 333 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικός για 333. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 ε, τζούρι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 335 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 336 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 337 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 338 υπέρ, κατά αποχές, έλεγχος ηλεκτρονικός παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τα υπόλοιπα καταπίπτουν μέχρι την 341. 341. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 3.42 υπέρ κατά να ελέγξουμε το 342 παρακαλώ να ψηφίσουμε και τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται 3-4-3 υπέρ. Έλεγχος για το 343 παρακαλώ. I'm closing the vote. Vote's closed. Uh, that's rejected. 17 to 20. Απορρίπτεται. 344 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 345 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας ελέγξουμε. Votes closed. Τέλος της πληροφορίας. Έγκρινεται. 3.46 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 346. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 3.47 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3.48 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική J υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική K και πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική M μη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική, ε, συγγνώμη, τροπολογία 432 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 433 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 404 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 435 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 436 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 437 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 438 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τζούρι 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 439 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 440 υπέρ κατά αποχές Διάφορες ενδιαφέρουσες χειρονομίες άκουσα. Είδα μάλλον. Ας ελέγξουμε παρακαλώ. Have τη voted? Votes closed. Πέρασε Απεριφθεί. Τώρα που πάμε στο επόμενο, Συμβαστική εν, νη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ζωμπόλ, μπερδεύτηκες. Εντάξει τώρα. Συμβαστική N νομίζω εγκρίνεται και έτσι πάμε στο δεύτερο τμήμα του καταλόγου των ψηφοφοριών. 466 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 447 υπέρ. Κατά αποχές. Να επαληθεύσουμε 447. Οπότε πάω να κάνω υποθέσεις, μπερδεύω, κάνω λάθος. Ας επαληθεύσουμε. Τρεις ακόμη πρόκειται να ψηφίσουν, ελπίζω. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Εγκρίνεται. 20 υπέρ, 16 κατά. 85 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 448. Α, όχι, έχει καταπέσει. Και αυτή έχει καταπέσει. Και πάμε στα 450 παρακαλώ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 451 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 452 είναι ρωσικού τύπου 453 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε παρακαλώ 453 Δύο ακόμη, ένας ακόμη, κλείνουμε το πετάλογο, απερίφθη. Συμβαστική O μικρόν, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική R ρο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 506 έχει αποσυρθεί και πάμε στην 507 υπέρ κατά αποχές. Να επαληθεύσουμε παρακαλώ. 507. Προσπαθώ να δω το ποτέ. Ανοίγουμε μάλλον ψηφοφορία. Για 507, πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 508 υπέρ. Α, είναι Είμαι καλός, αλλάζουμε σελίδα, ναι. Συμβαστική σίγμα S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 511 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε την 511. Παρακαλώ. Εψήφισαν όλοι, τη προφορίας, απερίφθη. 89 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 512 υπέρ κατά αποχές απερίφθη ελέγχουμε, ελέγχουμε 512 ηλεκτρονικός έλεγχος δύο ακόμα να ψηφίσουν πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 513 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 514 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 515 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 516 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 90 υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε παρακαλώ την 90 Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απερίφθη. 517 υπέρ. Κατά αποχές. Απερίφθη. 91 έχει αποσυρθεί. 518 υπέρ. Κατά αποχές. 518. Ψήφισαν όλοι. πέρας. Βγαίνουν τα ίδια νούμερα, αλλά με διαφορετικούς συνδυασμούς από ό,τι φαίνεται στην ψηφοφορία. 519 καταπίπτει, 520 παρακαλώ, υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 521 υπέρ, κατά επαληθεύουμε την 521. Μια ψήφος λείπει. Πέρας. Περίφθη. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 522 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 523 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 524 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 525 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 526 υπέρ κατά αποχές απερίφθε 527 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 528 υπέρ κατά αποχές, απεληθεύουμε την 528. Δύο ακόμα μένει να ψηφίσουν, παρακαλώ. Πέρας. Και εγκρίνεται. 529 κατά 530 παρακαλώ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 531 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 532 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 533 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 534 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, συμβαστική T υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική U υπέρ προφορική Προφορική. Υπάρχει διαφωνία για την προφορική. Επομένως πρώτα με την προφορική τροπολογία παρακαλώ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 566 υπέρ. Κατά αποχές. Επαληθεύουμε 566. Εγκρίνεται μάλλον, αλλά θα, το επαληθεύσουμε. Αν ψήφισαν όλοι, κλείνω την ψηφοφορία, όντως εγκρίνεται. 110. Δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. 111 υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται 567 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 568 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. 512 υπέρ κατά άποχες πρέπει να έχει εγκριθεί αλλά υπαλληθεύουμε. 112 ψήφισαν όλοι 14 της Επιτροπής των Νομικών Υποθέσεων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 570 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 571 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε την 571 παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Πέρας, εγκρίνεται. 572 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είπαμε να 16 τη Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 575 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 577 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 17 της επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 579 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται, 580 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 581 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε την 581 παρακαλώ ψήφισαν όλοι και εγκρίνεται 19 υπέρ, 17 κατά, άλλο συνδυασμό, άλλε ισορροπίε. 582 υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται, συμβιβιστική W παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται, 114 προφορική, τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 117 προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 156 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 114 υπέρ κατά αποχές απερίφθη ε, Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 508 ε, υπέρ κατά αποχές απερίφθη 589 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 590 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 591 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 118 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 119 υπέρ Κατά. Αποχές να επαληθεύσουμε την 119 παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εγκρίθηκε λοιπόν. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Και όντω εγκρίνεται. Τροπολογία πρώτη υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε 122 νομίζω ότι έχει εγκριθεί ψήφισαν όλοι πέρας λάθος έκανα απεριευθεί και άρα τα χέρια που σηκώνονται είναι άλλα από αυτά που πατάνε τα κουμπιά τα ίδια είναι όχι. 123 η ταυτόσημη. Την ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 2 έχει αποσυρθεί. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 128 υπέρ. Λάθος, έχει καταπέσει. 3. Έχει καταπέσει 129 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη 130 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 132 υπέρ. Κατά. Κατά. Να επαληθεύσουμε παρακαλώ. 132. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε, εγκρίνεται. Εκατόν τριάντα Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύμα σας παρακαλώ. 135. Ψήφισαν όλοι πέρας και εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Η 6 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ κατά. Αποχές επαληθεύουμε. 138. Εγκρίνεται. Πέρα Πέρας της Εγκρίθηκε. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συγγνώμη, συγγνώμη, μια στιγμή. Είπατε συμβιβαστική κάτι, ενώ εννοούσατε απλώς τροπολογία 8, σωστά, γιατί νομίζω ότι εκεί υπήρξε σύγχυση. Καλά, θα ξαναψεφίσουμε. Ναι, εννοούσα τροπολογία 8. Πράγματι. Θα ελέγξουμε υπέρ. Κατά. Αποχές ή ηλεκτρονικά. Πρόκειται για τη διαγραφή, έτσι. Τροπολογία 8. Ψηφίσατε πέρα της ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. 148 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίφθηκε. 149. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 150 είναι συμβατή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα το ελέγξουμε. Νομίζω ότι εγκρίθηκε, αλλά ας ελέγξουμε καλύτερα. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας, αλλά απορρίφθηκε. 19 κατά, 17 υπέρ. Συμβαστική Y υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 151 υπέρ, κατά, αποχές, δεν καταλαβαίνω από τα χέρια που σηκώνονται. Θα ελέγξουμε λοιπόν. 151. Ψηφίστε παρακαλώ. Άλλοι δύο πρέπει να ψηφίσουν. Πέρας φοφορίας. απορρίφθηκε. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 153 υπέρ. Κατά. Δεν καταλαβαίνω, θα ελέγξουμε. Δεν είδα τους σοσιαλιστές τι ψήφισαν. Ψηφίσατε όλοι υπέρ της φοφορίας, εγκρίθηκε. 154 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 155 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. 155. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ. Όχι, καταπίπτει. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Πρόεδρε, συγγνώμη που σας διακόπτω για την 158. Εδώ λέει σε μένα ότι δεν καλύπτεται. Α, ο δικός μου κατάλογος λέει ότι καλύπτεται, λέει πρόεδρος. Άλλαξε σήμερα το πρωί από ό,τι φαίνεται. Μια στιγμή. Υπάρχει κάπου πιο πέρα στον κατάλογο, σαν νέα. Θα την ψηφίσουμε δηλαδή, αλλά αργότερα στο νέο κατάλογο. Μην με ρωτήσετε γιατί, έτσι είναι. Τροπολόγια 10. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική Z. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, 158 για κάποιο λόγο. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε για την 158. Μπορείτε να ψηφίσετε. Στην καινούργια της θέση δεν ξέρω αν αυτό αλλάζει κάτι. Είναι πάντα στην ατυλογική σκέψη 18α. Τέλος πάντων. Πέρα στις φοφορίες απορρίφθηκε. Με δύο ψήφους διαφορά. 160 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 12 έχει αποσυρθεί. 163 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε 163. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. 21 ψήφοι υπέρ. Εγκρίνεται. 164 υπέρ. Παρακαλώ, Σόφη. Μπορεί να φταίει ο δικός μου κατάλογος ψηφοφορίας, αλλά τι έγινε με την 159. Δεν καλύπτεται από το συμβασμό, τουλάχιστον στον κατάλογο που έχω εγώ. Πρόεδρος, από ό,τι φαίνεται καλύπτεται από τη συμβιβαστική Z. Σήμερα το πρωί άλλαξαν τα πράγματα. Ωραία, εγώ έχω την παλιότερη εκδοχή τότε, λέει η κυρία Ινφετφέλτ. Πρόεδρος, ωραία, συνεχίζουμε. 164. Έτσι, εκεί ήμασταν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. 167. Ψηφίστε. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Άλλοι δύο πρέπει να ψηφίσουν. Πέρα τη ψηφοφορία. Όχι, απορρίφθηκε. Καλά, δεν θα ξανακάνω προβλέψεις. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. 169 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 170 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 171 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 172 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 173 υπέρ, κατά, ελέγξουμε καλύτερα. 173. Πέρας της φοφορίας. Άλλος ένας Πέρας. Εγκρίθηκε με μία ψήφο διαφορά. 173 δεν ήταν αυτή, ναι, εγκρίθηκε. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 177 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 178 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 179 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 181 υπέρ, κατά αποχές θα ελέγξουμε 181. Ψηφίστε. 181 πέρα στις φοφορίες εγκρίνεται. 180 καταπίπτει. 182 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 185 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 184 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 186 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Αποσύρθηκε 18, 187 υπέρ, κατά αποχές θα ελέγξουμε 187. Μπορείτε να ψηφίσετε. Άλλος ένας, πέρας της φοφορίας. Απορρίφθηκε. 17-19. 188 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 189 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 190 καταπίπτει. 191 τώρα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 194 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε 194 ψηφίστε άλλος ένας Πέρα της φοφορίες. Εγκρίνεται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 196 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 197 υπέρ. Κατά. θα ελέγξουμε. 197. Εδώ βλέπω διπλά και τριπλά, λέει η πρόεδρος. Ψηφίσατε όλοι, εγκρίθηκε 19-17 το αποτέλεσμα. 201 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 202 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 203 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 204 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 205 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 205 να ελέγξουμε καλύτερα. Εντάξει, γιατί μπορεί να κάνω και λάθος. Μπορεί. Πέρα στις φοφορίες. Δίκιο είχα. Όχι, λάθος είχα. Εγκρίνεται τελικά. 206. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. 206. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 207 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 208 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 209 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 210 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 211 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 212 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 213 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 214 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά τώρα θα ψηφίσουμε το τροποποιημένο κείμενο. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψήφισατε όλοι. 36 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά και καμία αποχή. Το νομοθετικό ψήφισμα τώρα. Ψηφίζουμε. Πάλι με 36 ψήφους υπέρ, καμία ψήφο κατά και καμία αποχή. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ και θα ήθελα μόνο να Ευχαριστήσω τους σκιώδες εισηγητές. Υπάρχει μια βούληση ώστε αυτή η ψηφοφορία να περάσει άμεσα στην Ολομέλεια και αν είναι δυνατόν να επιτύχουμε θετική ψηφοφορία σήμερα στην Επιτροπή. Γι' αυτό Προτείνω να μην ε, ψηφίσουμε για έναρξη διαπραγματεύσεων, αλλά να πάμε κατευθείαν στην Ολομέλεια. Τέλο, θα ήθελα να πω δύο λόγια, όλο ιδιαίτερο, για όλου του τεχνικού ε, βοηθού τη Επιτροπή μα που μα βοήθησαν. Θα ήθελα επίση να σα δώσω μία, να πω δύο λόγια μάλλον και να ευχαριστήσω την Μαφάλδα που, για την ε, βοήθεια που μα έδωσε την Όδη, τη Σοφή, τον Ζανπόλ, τον Γιούργεν και όλους όσους βοήθησαν για να πετύχουμε αυτά τα αποτελέσματα που σίγουρα δεν θα είχαν καταστεί δυνατά χωρίς τη βοήθειά σας. Και ε, ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. I think we may have had some uh, differences in the interpretations going on there. Ε, υπάρχουν τώρα εδώ κάποιες διαφορέ ερμηνείες. Ο εισηγητής λοιπόν λέει ότι δεν επιθυμεί να μπει σε διαπραγματεύσεις σε αυτή τη φάση. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε τη διαπραγματευτική αυτή εντολή. Πάμε κατευθείαν στην Ολομέλεια όπου βεβαίως μπορούμε να επιλέξουμε να, να στείλουμε την τελική ψηφοφορία ώστε να γίνουν οι διαπραγματεύσεις. Αυτό λοιπόν θα πάει στην Ολομέλεια. Εντάξει, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε για την έναρξη των διαπραγματεύσεων, γιατί δεν τίθεται το ζήτημα. Οπότε λοιπόν προχωράμε στην έκθεση του Πάμπλο. <laughs> Ah. If you Αν ψηφίζετε όλο το ίδιο όλη την ώρα, θα πάμε και πιο γρήγορα. Λοιπόν, συμβιβαστική α, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, μάλλον όχι δεν εγκρίνεται, ελέγχουμε. Okay, we're down to 33 people as well. We're closing the vote. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με πολλούς που δεν είδα να ψηφίζουν υπέρ. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξω γιατί έχουν φύγει κάποιοι και δεν ξέρω τώρα πώς βγαίνουν τα νούμερα. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 18 προς 16. Τροπολογία 5 υπέρ. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχές. Να ελέγξουμε την τροπολογία 5. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με μία ψήφο διαφορά. Αχ, δύσκολη ζωή μου κάνατε σήμερα. Ε, 98 υπέρ κατά. Ας ελέγξουμε για την 98. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Two more to vote, one more to vote, one more to vote. If you're not voting, I'm closing. Thank you. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μία ψήφο. 104. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 105. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 106. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 107. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, να ελέγξουμε την 107. Voted, votes closed. Τέλος της ψηφοφορίας και εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική β με προφορική τροπολογία την οποία πρέπει να διαβάσω λέει θα διαβάσω όλο αυτό το κομμάτι δηλαδή λέει έχει δύο νέες λέξεις οι νέε λέξει είναι immediately, άμεσα και έχει καθαριστεί. Η συναλλαγή χρεωστική μέσω κάρτα σημαίνει μία ε, πληρωμή που βασίζεται σε κάρτα και συνδέεται με έναν τρέχοντα ε, λογαριασμό ή λογαριασμό καταθέσεων στον οποίο ε, χρεώνεται η συναλλαγή άμεσα αφού έχει εκαθαριστεί. Ενώ μια συναλλαγή με μια προπληρωμένη κάρτα είναι χρεωστική συναλλαγή με κάρτα. Αυτά λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κοιτάξτε, εκεί λίγο φωνάζετε με το τηλέφωνο και με ενοχλείτε, με μπερδεύομαι. Συμβιβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εγκρίνεται 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 130 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οτροπολογία 8 υπέρ κατά Αποχές. Ελέγχουμε. Για την 8. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικός. Every voted, votes closed. Τέλος ψηφοφορίας. Έγκρινεται. 17 προς 15. Ε, τροπολογία 9, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 9. Κανείς δεν ψη... Ε, ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας καταπιπτεί, απορρίπτεται δηλαδή. 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 139 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 139 Απορρίπτεται. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 140 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 141 υπέρ, κατά αποχές να ελέγξουμε την 141. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές α, ελεγχός ηλεκτρονικός. Καταπίπτει. Ήμκο 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 145 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ΙΜΚΟ 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 148 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ γιατί κάποια χέρια δεν τα είδα Ξέρω ότι καλύτερα είναι να κουβεντιάζει κανείς, αλλά πρέπει να ελέγξουμε ωστόσο. Απορρίφθηκε 149 ε, υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται 150 υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται 153 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά θα ελέγξουμε για τη 10 απορρίπτεται 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική D πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στην συμβιβαστική ε Ευτυχώ πηδάμε έτσι και μερικέ σελίδε. Συμβιβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.37 2.37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.39 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε τη 239 Ε, εγκρίνεται. 240 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 241 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικός τέλος πληροφορίας. απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξω πάλι Δύο ακόμα μένουν να ψηφίσουν. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δύο υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξω το 244. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 17 προς 15. 18 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε... Καταπίπτει. Συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 250 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 26. Α, κουραστική η γραμματεία και μου πελάθο. Σύμκο 26. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 251 υπέρ. Κατά αποχές Καλύτερα να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας, απορρίπτεται με μία ψήφο. Διαφορά. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 254 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. 255 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 261 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά 261 Εγκρίνεται υπέρ. 263 ε, υπέρ κατά αποχές απερίφθη 264 υπέρ κατά αποχές πρέπει να επαληθέσουμε τη 264 264 ψήφισαν όλοι εγκρίνεται 265 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 266 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 267 όχι καταπέπτει 268 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 269 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 271 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 270 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβαστική FA πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε την 21 Ψηφίσατε όλοι. Απεριφθεί 29 της ΕΜΚΟ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 276 υπέρ. Κατά αποχές απεριφθεί. 22 υπέρ. Κατά αποχές επαληθεύονται 22. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφορίας. Απεριφθεί. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές απεριφθεί. Και επαληθεύω. Απερίφθη. δύο ψήφου διαφορά. 283 επομένω. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απεριφθεί 284 υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε τη 284. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε. Απεριφθεί. 25 υπέρ. Κατά. Θα την επαληθεύσουμε. 25. Την 25 παρουσιάζουμε. Απερίφθη. 291. Υπέρ. Κατά. Αποφε, αποχές. Απερίφθη. 292. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Συμβαστική G, ζήτα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 298 υπέρ κατά αποχές. Απερίφθη 299 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 300 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 31 της ΣΥΜΚΟ υπέρ κατά 31 Πέρασε. Απερίφθη. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 301 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 8 συμβαστική, H συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 34 τη ΣΥΜΚΟ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 305 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 τη ΣΥΜΚΟ έχει καταπέσει μάλιστα 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 306 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 306 υπέρ 316 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 308 υπέρ κατά εποχές απερίφθη 307 υπέρ κατά επαληθεύω 307 ψήφισαν όλοι πέρας κατά πίπτη 16 απερίφθη μάλλον 16 υπέρ και 16 κατά συμβαστική ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική K τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά Αποχές επαληθεύουμε. Εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Γεμικό 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική L, λάμδα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. M, μη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική N, νη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. O όμικρον, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. P υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, Επαληθεύουμε. Ψήφισαν όλοι. Εγκρίνατε. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη νομίζω, αλλά σε παρηθεύσουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 66 υπέρ. Κατά αποχές, επαληθεύω, αν και νομίζω ότι έχει εγκριθεί. Οπότε θα αποδειχθεί πως έχω άδικο, αλλιώς δεν θα χρειάζεται να επαληθεύσω. Ψήφισε όλοι, όλια, είχα και δίκιο λοιπόν, 15 κατά, 17 υπέρ, συμβαστική Q υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 7 τη ΣΥΜΚΟ υπέρ, κατά αποχές απερίφθη, 2 υπέρ, κατά αποχές. Επαληθεύω την υπαριθμόν δύο τροπολογία. η οποία καταπερίφθη απερίφθη 16 ψήφι κατά, 16 ψήφι υπέρ. 70 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 71 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 72 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε την 72 παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. Απερίφθη 16 ψήφους κατά, 73 υπέρ, κατά. Αποχές απερίφθη 3 υπέρ κατά, επαληθεύουμε την 3. Απερίφθη. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 8 τη σημικό υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Συμβαστική R, ρο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 83, υπέρ, κατά. Α, δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, παρακαλώ να επαληθεύσουμε. 83. Εγκρίνεται. 9 τη ΣΥΜΚΟ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, 84 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. Ηλεκτρονικά το κείμενο όπως τοποποιήθηκε. Λείπουν ακόμα δύο ψήφοι, πέρας ψηφοφορίας, 26 υπέρ. 5 αποχές και χωρίς ψήφους κατά. Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, παρακαλώ. Ακόμα λείπει μία ψήφος. Πέρας. 25 υπέρ. 3 κατά, 2 αποχές. Sharon, first of all, I would like to... Σέρον, ευχαριστώ πολύ. Θα να ευχαριστήσω τώρα από τον φίλο Τιέγκο, την ε, βοηθό του Μαθάλτα, το δικό μου το γραφείο με το Σαλβαδόρ ιδιαίτερος και βέβαια και τη γραμματεία της Επιτροπής και ως, όπως πάντα τους σκιώδεις συγκητές με τους οποίους ήταν τιμή και χαρά στη συνεργασία όλους τους ε, αναφέρω όλους έναν έναν και προτείνω να προχωρήσει το θέμα αυτό στην Ολομέλεια ώστε να ενισχύσουμε το ρόλο του Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε πολύ. Θα πάει στην Ολομέλεια αυτόματα. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε εντολή για τις διαπραγματεύσεις. Και τελική ψηφοφορία θα εξαρτηθεί από το τι θα αποφασίσουμε τότε. Συνεχίζουμε και περνάμε σε κάτι διαφορετικό. Ψηφίζουμε γνωμοδοτήσεις όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών πρώτα. Απαλλαγές. Συμβαστική Α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. δύο Υπέρ Κατά. Α, δεν ξέρω εδώ ποιο είναι το αποτέλεσμα. Μπέρδεμα. Λοιπόν, ψηφίζουμε την τροπολογία 2. Εδώ βλέπω πολύ κινητικότητα στην αίθουσα. ρε, ποια από τις τρεις ψηφίζουμε, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει ποια από τις τρεις γνωμοδοτήσεις. Μα το είπα, λέει η Πρόεδρος. Για λίγο ηρεμία. Ψηφίζουμε. Αϊόπα. Για ποια αρχή να μας πείτε, για ποια αρχή από όλες ψηφίζουμε. Ωραία, ξανά ψηφίζουμε την απαλλαγή της αρχής ασφαλίσεων. Δεν είναι εύκολο όντως να καταλάβει κανείς. Έχετε όλοι το αιώπα επειδή υπήρξε σύγχυση. Αρχίζουμε και πάλι λοιπόν. Συμβαστική Α. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική Σ, γάμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική δέλτα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική ε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Άλλος ένας, πέρα της φοφορίας. 24 υπέρ, 3 αποχές, καμία ψήφος κατά. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στην ΕΣΜΑ. Συμβαστική Α. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική Β. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική γάμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο 6 παράγραφος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. «24 ψήφοι υπέρ, τρεις αποχές, καμία ψήφος κατά. Και έτσι τώρα φτάνουμε στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Έχετε τον κατάλογό σας, συμβαστική α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική β υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αρχική παράγραφος 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική γ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίν... απορρίπτεται. Συμβαστική δέλτα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική ε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά παρακαλώ. 22 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά και 3 αποχές. Ευχαριστώ. Σας υπενθυμίζω πρώτα απ' όλα ότι θα ψηφίσουμε με τη ΛΥΜΠΕ στις 12.30. Δύο όροφοι πιο πάνω δηλαδή. Να έχετε τις κάρτες σας μαζί και η επόμενη συνεδρίαση ΕΚΟΝ είναι τη Δευτέρα στις 7.30. 4 και είναι στις 12.30 τώρα που θα ψηφίσουμε με την ΛΥΜΠ, έτσι, στις 12.30. Και έλεγα ότι συνεδριάζουμε και πάλι τη Δευτέρα στο Στρασβούργο στις 7.30 μετά μεσημβρίας. Ευχαριστώ πολύ και για τη βοήθεια στη ψηφοφορία.